Iniziamo. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν έρθει ακόμα οι περισσότεροι συναδελφοί, αλλά ο χρόνος περνάει και στις 4.30 πρέπει να τελειώσει το εργαστήριο, διότι όπως θα θυμάστε θα έρθει το ελεγκτικό συνέδριο, πιο συγκεκριμένα ο εισηγητής ο κύριος Κρετών για την ε, έκθεση για τις προτάσεις μεταρρύθμισης και θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε χωρίς περαιτέρω καθιστήριο, πολύ σημαντικό εργαστήριο Αγαπητοί συνάδελφοι, η αδυναμία των γεωργών για την διατροφική αλυσίδα είναι κάτι το οποίο μας αποσχάλεσε προσφάτως στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 19 ε, Ιανουαρίου του 2012 επί τη βάση της έκθεσης της Επιτροπής Γεωργίας για την ε, αλυσίδα διανομής ε, της γεωργικής παραγωγής, τη δομή και τις επιπτώσεις. Και εκεί διαπιστώσαμε ότι υπάρχει αύξηση της αβεβαιότητας ε, και της ανασφάλειας των γεωργικών προϊόντων και των μακροπρόθεσμων επενδύσεων των γεωργών. Και επίσης ε, διαπιστώσαμε ότι οι πιο αυξημένες ε, τιμές των τροφίμων για τους καταναλωτές δεν σημαίνουν απαραίτητο ότι είναι πιο αυξημένα και τα εισοδήματα των γεωργών. Και σε αυτό το πλαίσιο βεβαίω, στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της κοινή γεωργικής πολιτικής, περνάμε σε αυτό το πλαίσιο ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τους ειδικούς κανόνες για την τροφική αλυσίδα στη νέα ΚΑΠ. Καλωσορίζω λοιπόν εδώ τους εμπειρογνώμονές μας, τον, την καθηγήτρια Κατρίν Τελκόντ του Πανεπιστήμιου της Νάντης, τον καθηγητή Αντώνιο Τζαναρέλη από το Πανεπιστήμιο του Μπάρι και και τον κύριο Μποντιγκέλ από το Γαλλικό ε, Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας ε, στην Άντι. Θα δώσω κατευθείαν το λόγο στην ε, καθηγήτρια Ντελκόντ. Έχετε όλοι μαζί ένα τέταρτο με 20 λεπτά για την παρουσίαση της μελέτης. Στη συνέχεια θα ξεκινήσει η συζήτηση και κατόπιν θα σας δώσω και πάλι το λόγο για να απαντήσετε στις ερωτήσεις που θα σας διατυπώσουν οι συνάδελφοι. Παρακαλώ κύριε Ντελκόντ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, το θέμα της έκθεσης αυτής είναι να αναλύσει το ουσιαστικό δίκαιο του ανταγωνισμού και την εφαρμογή του στη Γεωργία. Κατόπιν αναλύει την πρόταση της νέας ενιαίας κοινής οργάνωσης αγοράς και συγκεκριμένα τις διατάξεις που άπτονται την οργάνωση των διαφόρων κλάδων και το δικαίωμα του ανταγωνισμού. Τέλος, προτείνει κάποιες συστάσεις, συστάσεις ε, που λαμβάνουν υπόψη την ιδιαιτερότητα της γεωργίας και την ανάγκη επανισορρόπησης της αλυσίδας ε, τροφίμων. Ποιο είναι το σημείο αφετηρίας λοιπόν της ε, μελέτης αυτής. Φυσικά σημείο αφετηρίας είναι το άρθρο 48 της συνθήκης για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει ότι οι κανόνες που άπτονται του ανταγωνισμού δεν εφαρμόζονται στην παραγωγή και στο εμπόριο των γεωργικών προϊόντων ε, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1 παρά μόνο στο, στο μέτρο που προσδιορίζεται κάτι τέτοιο από το Συμβούλιο στη συνθήκη της ε, Ρώμης και ε, όπως με τη νέα συνθήκη καθορίζεται από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Το 40, άρθρο 42 μάλιστα ε, αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα της γεωργίας και την κοινωνική λειτουργία της κοινή ε, γεωργικής πολιτικής. Αυτή λοιπόν η κοινωνική λειτουργία της κοινή γεωργικής πολιτικής θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εφαρμογή των ε, κανόνων ανταγωνισμού. Πώς εφαρμόστηκε λοιπόν, ενσωματώθηκε και ερμηνεύτηκε η αρχή αυτή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού και ως προς τη Γεωργία. Έχουμε καταρχήν τον κανονισμό 2662 που αφορούσε την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στη Γεωργία. Ο κανονισμός αυτός 26 του 1962 ανέτρεψε την αρχική φιλοσοφία του άρθρου 42 γιατί σας υπενθυμίζω ότι το άρθρο 42 προέβλεπε ότι οι κανόνες ανταγωνισμού δεν εφαρμόζονται παρά μόνο στο μέτρο που καθορίζεται κάτι τέτοιο από το Συμβούλιο. Ενώ ο κανονισμός του 1962, υπαριθμόν 26, ανατρέπει αυτή την αρχική φιλοσοφία, προσδιορίζοντας ότι οι αρχές του κανόνων ανταγωνισμού εφαρμόζονται και στη γεωργία και μόνο κάποιες εξαιρέσεις αναγνωρίζονται όπως αναφέρονται στον κανονισμό. Μόνο μερικές εξαιρέσεις επιτρέπονται. Αυτή η αντιστροφή της ε, προσέγγισης, ε, αυτή η ανατροπή της αρχικής φιλοσοφίας περιλαμβάνεται όχι μόνο στον κανονισμό 26 του 62, αλλά και στον κανονισμό 1144 του 86, αλλά και στον ισχύοντα κανονισμό για την ενία ΚΟΑ και επίσης ε, την ερμηνεία και την εφαρμογή των εξαιρέσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εν κατακλείδη λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι σημείο αφετηρίας ήταν ε, μια ε, εφαρμογή που καθορίζεται από το Συμβούλιο και ε, στο ισχύον ουσιαστικό δίκαιο από το 1962 έχουμε μια ανατροπή αυτής της φιλοσοφίας γιατί καταρχήν εφαρμόζουμε και στη γεωργία τους κανόνες ανταγωνισμού με ορισμένες μόνο εξαιρέσεις και αυτές οι εξαιρέσεις περιορίζονται στο, στα δικαιώματα των συμφωνιών. Τρία είναι τα είδη των εξαιρέσεων που επιτρέπονται. Καταρχήν, οι εξαιρέσεις που αφορούν κάποιες πρακτικές των εθνικών οργανώσεων αγοράς. Αυτή η εξαίρεση θα καταργηθεί γιατί οι εθνικές οργανώσεις αγοράς επίσης θα καταργηθούν. Μια δεύτερη εξαίρεση αφορά τις συμφωνίες που είναι απαραίτητες για να υλοποιηθούν οι στόχοι της κοινή γεωργικής πολιτικής. Και τρίτο είδος εξαιρέσεων που επιτρέπονται είναι οι εξαιρέσεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 177 της κοινή ΚΟΑ και που αφορούν τις, ε, ε, τα interprofession, τις διακλαδικές οργανώσεις. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού από το 1962 φαίνεται ότι υπερισχύει η πολιτική ανταγωνισμού επί της πολιτικής γεωργίας και το ιδιαίτερο καθεστώς ε, που ε, ίσχυε μόνο για την ε, γεωργία πριν το 1962 έχει περιοριστεί. Πολλό δε μάλλον που η εφαρμογή αυτών των κανόνων, η ερμηνεία αυτών των κανόνων από την Επιτροπή και το ΔΕΚ είναι πολύ συσταλτική και de facto έχει διαμορφωθεί μια λειτουργική ιεραρχία μεταξύ της πολιτικής ανταγωνισμού και της κοινή γεωργικής πολιτικής. Μια η ιεραρχία που απουσιάζει πλήρως από τα κείμενα της συνθήκης. Ποιο είναι λοιπόν το πλαίσιο που προτείνεται στη νέα πρόταση 126 για την κοινή οργάνωση αγοράς. Το γενικό πλαίσιο της πρότασης προβλέπει ε, διεύρυνση των κανόνων της, των ισχυωσών ΚΟΑ, οποροκυπευτικά, ε, καπνός και άλλα και για ορισμένα μέτρα του γάλακτος να τα επεκτείνει σε όλους τους τομείς. Και επεκτείνει κυρίως τους κανόνες που αφορούν την αναγνώριση των επαγγελματικών οργανώσεων, τους κανόνες που αφορούν τις συμφωνίες οργανώσεων ε, παραγωγών ή των διεπαγγελματικών οργανώσεων και το θέμα της ε, σύναψης ε, συμβολέων ε, μεταξύ των διαφόρων παραγωγών, την ενοχική δηλαδή πτυχή. Τώρα, μερικές ε, παρατηρήσεις για τις, οργανώσεις, τις επαγγελματικές οργανώσεις. Έχουμε το άρθρο 120, 100, της συνθήκης, παράγραφος Δέλτα, που περιλαμβάνει μία νέα καινοτομία και που προβλέπει απαγόρευση της δεσπόζουσας θέσης, μια απαγόρευση που δεν υπάρχει στο κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμού. Το άρθρο 106 Δέλτα απαγορεύει στις οργανώσεις να δημιουργήσουν δεσπόζουσα θέση. Ενώ το κοινοτικό δίκαιο επιβάλλει κυρώσεις μόνο στην κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης. Δεν εμποδίζει τη διαμόρφωση δεσπόζουσας θέσης. Έχουμε λοιπόν μια διάταξη που ε, αντιβαίνει στο ισχύον δίκαιο του ανταγωνισμού. Και μάλιστα το κείμενο αυτό, 106 Δέλτα, αντιβαίνει και στο άρθρο 111 της ίδιας πρότασης. Γιατί για να θεωρηθεί ως αντιπροσωπευτική, μία οργάνωση οφείλει να έχει δεσπόζουσα θέση. Αλλιώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αντιπροσωπευτική. Και αυτή η διάταξη αντιβαίνει και με τους στόχους που περιλαμβάνονται στην αιτιολογική σκέψη 85 του κειμένου, ε, η αιτιολογική σκέψη μιλάει για ενίσχυση της συγκέντρωσης των διαφορών φορέων και ενίσχυση της διαπραγματευτικής τους ισχύω απέναντι στους οικονομικούς τους εταίρους. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ενοχική πτύχη, το ενοχικό σκέλος, έχουμε τον κανονισμό 261 του 2012 που ε, επιβάλλει την υποχρέωση γραπτής σύμβασης για κάθε παράδοση γάλακτος. Και νομίζω ότι και η διάταξη αυτή έχει σχέση με τους κανόνες ανταγωνισμού. Οι κανόνες ανταγωνισμού σε καμία περίπτωση δεν τροποποιούν την αρχή με βάση την οποία οι κανόνες ανταγωνισμού ισχύουν και για τη γεωργία. Απλώς μιλάει για την, επαβεβαιώνει την αρχή τη, της εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού και αναφέρει τις ίδιες εξαιρέσεις με μία διαφορά την ε, εισαγωγή αυτής της περίφημης απαγόρευσης ε, κατοχής δεσπόζουσας θέσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους κανόνες ανταγωνισμού που ισχύουν για τις οριζόντιες συμφωνίες, δηλαδή τις συμφωνίες των παραγωγών, έχουμε μία επέκταση των μέχρι τώρα διατάξεων του συστικού δικαίου έχουμε διατήρηση της ε, ε, απαγόρευσης των ρητρών για τις τιμές και έχουμε την μείζωνα καινοτομία που είναι ε, η απαγόρευση της κατοχής δεσπόσας θέσης. Ό,τι αφορά τις επαγγελματικές οργανώσεις, δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη καινοτομία στο κείμενο, παρά μόνο την επέκταση της προηγούμενης εξαίρεσης που στο παρελθόν αφορούσε μόνο τα απορροκυπευτικά προϊόντα. Σε ό,τι φορά τώρα τις διατάξεις του ανταγωνισμού, θα λέγαμε ότι οι νέες αλλαγές είναι ίσονο σημασία παρά τους ε, ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους που περιλαμβάνονται στις αιτιολογικές σκέψεις. Δηλαδή, στόχος είναι η ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης ε, απέναντι στους οικονομικούς εταίρους και επίση θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτέ οι νομικέ αλλαγέ, αυτέ οι ένομε αλλαγέ δημιουργούν κάποια ερωτηματικά σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των προτινόμενων διατάξεων σε σχέση με τους στόχους που έχουμε να υλοποιήσουμε. Τέλος, αυτή η πρόταση θα μπορούσαμε να πούμε ότι επιβεβαιώνει την υπεροχή της πολιτικής ανταγωνισμού επί της, πολιτικής, της γεωργικής πολιτικής. Τι προτείνουμε. Εμείς προσπαθήσαμε να υποβάλουμε κάποιες συστάσεις που ε, στόχο έχουν να μας βοηθήσουν στην υλοποίηση των ακόλουθων στόχων. Καταρχήν, σωρόπιση της ε, αλυσίδας τροφίμων και ε, επαναφορά του ρυθμιστικού ρόλου της γεωργίας, του ρυθμιστικού πλαισίου της γεωργίας, προκειμένου να ληφθούν υπόψη ιδιαιτερότητες του γεωργικού κλάδου. Άλλος στόχος είναι να επιτρέψουμε στους γεωργούς και στις επαγγελματικές οργανώσεις να γίνουν πραγματικοί φορείς και παράγοντες της ρύθμισης. Και τέλος, να επιτρέψουμε στους στόχους του άρθρου 39, τους στόχους δηλαδή της κοινής γεωργικής πολιτικής, να, ε, να αναλυθούν υπό το φως της ε, μέχρι τώρα εμπειρία μας, ε, μέχρι τώρα εμπειρίας μας, αλλά και ε, υπό το πρίσμα της αναμενόμενης μεταρρύθμισης της ΚΑΠ και μάλιστα θέλοντας να βελτιώσουμε την ε, συνοχή και τη συμβατότητα των κειμένων που ισχύουν για τη γεωργία και να θέλουμε να βελτιώσουμε και την αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με την ερμηνεία που δίνουν η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οπότε η μελέτη αυτή μας κάνει μια επισκόπηση της σημερινής κατάστασης του ουσιαστικού δικαίου και μας προτείνει κάποιες συστάσεις για να ισχυθεί η αποτελεσματικότητα των εξαιρέσεων. Εγώ θα επικεντρωθώ στις βασικές συστάσεις, γιατί υποβάλαμε αρκετές συστάσεις. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τους κανόνες ανταγωνισμού. Ε, ως προς το άρθρο 144 και τις ε, εξαιρέσεις ε, για τους στόχους της ΚΑΠ και τις οριζόντιες οργανώσεις, τις οργανώσεις ε, παραγωγών, προτείνουμε ένα τεκμήριο συμβατότητας των συμφωνιών με το δίκαιο ανταγωνισμού. Με άλλα λόγια, οι συμφωνίες και οι πρακτικές των παραγωγών και των οργανώσεών τους θα πρέπει να θεωρηθούν, να, να τεκμέρονται ότι υλοποιούν τους στόχους της κοινή γεωρικής πολιτικής. Οπότε αντιστρέφουμε το βάρος απόδειξης και εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποδείξει ότι αυτές οι συμφωνίες των παραγωγών ή των οργανώσεών τους αντιβαίνουν στην υλοποίηση των στόχων της ΚΑΠ. Δεύτερη πρόταση για το άρθρο 144 είναι η κατάργηση της απαγόρευσης κατοχής δεσπόζουσας θέσης για αυτές τις οργανώσεις παραγωγών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δύο επαγγελματικέ οργανώσεις, δεν προτείναμε σημαντικές ε, αλλαγές στο κείμενο, αλλά προβληματιστήκαμε ως προς την ανάγκη να ε, κρατήσουμε αυτή την ε, προηγούμενη κοινοποίηση των συμφωνιών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάλαμε αυτό το ερωτηματικό. Αν διατηρηθεί αυτή η προηγούμενη κοινοποίηση προς την Επιτροπή, θα πρέπει ταυτόχρονα να θεσπιστούν κανονισμοί εξαίρεση ανακατηγορία, προκειμένου να ε, περιληφθούν σε κατάλογο οι συμφωνίες, οι ρήτρε ε, που θεωρούνται συμβατές με το δίκαιο του ανταγωνισμού από τη στιγμή που θα περιληφθεί ένα τέτοιο κατάλογο, είτε, στη βασική, είτε στη βασική πράξη, είτε σε ένα κανονισμό με εξαιρέσει, τότε ε, η προειδοποίηση γίνεται άνευ προηγουμένου. Η προηγούμενη προειδοποίηση. Γιατί σε τέτοια περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα προβούν σε μια αυτοαξιολόγηση των συμφωνιών του με βάση το δίκαιο ανταγωνισμού. Τώρα, αν θεσπιστεί ένα κανονισμό εξαιρέσεων ανακατηγορία για τις διαπαγγελματικές οργανώσεις, είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι ένας τέτοιος κανονισμός εξαιρέσεων θα ε, άπτονταν των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου με βάση το άρθρο 42 της Συνθήκης. Μια και θα πρέπει να καθοριστεί σε ποιο μέτρο, σε ποιο βαθμό οι κανόνες ε, ανταγωνισμού, το δίκαιο ανταγωνισμού ισχύει για τη γεωργία. Γιατί αυτό είναι το περιεχόμενο του άρθρου 42 της Συνθήκης. Τέλο, ό,τι αφορά και πάλι τις διαπαγγελματικέ οργανώσεις, κρίναμε σκόπιμο να προσθέσουμε μία διάταξη που ε, επιτρέπει τη λήψη υπόψη των ε, κατεπηγουσών καταστάσεων, των περιπτώσεων κρίσης, ώστε να είναι δυνατή η άμεση αντίδραση και αντιμετώπιση των κρίσεων. Πρόσφατα, το περασμένο καλοκαίρι, είχαμε παρόμοια κρίση στον τομέα των απορροκυπευτικών. Μία άλλη σύσταση που κατά τη γνώμη μας είναι θεμελιώδους σημασία, στα πλαίσια των άρθρων 144 και 145, των εφαρμοστέων δηλαδή ε, κανόνων ανταγωνισμού για της συμφωνίες, είναι η κατάργηση της ε, απαγόρευσης σύναψης συμφωνιών για τον ορισμό τιμής. Η απαγόρευση ρήτρας καθορισμού τιμής είναι ευνόητη γιατί έχουμε μια κοινή γεωργική πολιτική. Ήταν ευνοήτη όταν είχαμε μια κοινή γεωργική πολιτική που στηριζόταν σε διοικητικέ τιμέ. Από τη στιγμή όμω που οι διοικητικέ τιμέ, παρόλο που υπάρχουν ακόμη, δεν επιτελούν όμω την ίδια λειτουργία, δεν έχουν δηλαδή αυτή τη λειτουργία του προσανατολισμού των τιμών τη αγορά, είναι πλέον περιττό, για να μην πω αντιφατικό, να παραμείνει ενισχύ η απαγόρευση ε, των ρητρών ε, ορισμού τιμών, καθορισμού των τιμών. Άσχετα αν πρόκειται για οριζόντιες ε, συμφωνίες μεταξύ παραγών ή κάθετες μεταξύ οργανώσεων παραγωγών, πιστεύω ότι μπορούμε να καταργήσουμε αυτή την απαγόρευση της ρήτρα καθορισμού των τιμών. Άλλωστε το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι πολύ πιο αυστηρό στην περίπτωση αυτή ως προς το, από το αμερικανικό δίκαιο. Συγγνώμη. Και με την ίδια λογική θα πρέπει, θα, καλό θα ήταν για να είμαστε συνεπείς να καταργήσουμε και την απαγόρευση ε, το, της κατοχής της πόσας θέσης. Τέλος και θα ολοκληρώσω γιατί εξέλιξε το χρόνο μου. Τα άρθρα και 105 για το γάλα εμπίπτουν μέσω του άρθρου 185 του κανονισμού του 2012 στο ε, ουσιαστικό δίκαιο. Θα πρέπει όμως να δούμε ποια είναι η εμβέλεια αυτής της υποχρέωσης γραπτών συμβάσεων. Στο μέτρο που ο στόχος είναι η εξασφάλιση της διαφάνειας των διαπραγματεύσεων, στο μέτρο που ο στόχος της υποχρέωσης ε, σύναψης γραπτών συμβάσεων είναι η επανισορρόπηση των ενοχικών σχέσεων, θα ήταν λογικό η υποχρέωση αυτή να επεκταθεί σε όλους τους τομείς. Γιατί η διαφάνεια και η επανισορρόπηση των ενοχικών σχέσεων δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στον τομέα το γαλακτοκομικό. Κατά συνέπεια, σκόπιμο θα ήταν να εξετάσουμε την θέσπισε ένα κανόνα που επιβάλλει υποχρέωση σύναψη γραπτών συμβάσεων για όλους τους κλάδους, για όλους τους τομείς. Εν κατακλείδη, θα μπορούσαμε να πούμε για τη μελέτη αυτή ότι η πολιτική ανταγωνισμού, όπως εφαρμόζεται στη Γεωργία, θα έπρεπε να αντανακλά τις ιδιαιτερότητες αυτού του κλάδου της Γεωργίας και όχι να προσπαθεί να τις εξουδετερώσει ή να τις σβήσει. Μόνο μια νομοθετική δράση θα μπορούσε να προωθήσει και να δικαιολογήσει μια τροποποίηση της εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού στην παραγωγή και εμπορία γεωργικών προϊόντων. Και μόνο μια νομοθετική αλλαγή, μια νομοθετική μεταρρύθμιση θα δικαιολογούσε αλλαγή της ερμηνείας των εξαιρέσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Συμπερασματικά λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι για να έχει νόημα ή να αποκαταστήσουμε την αρχική σημασία του άρθρου 42 και για να ξαναδώσουμε ε, την, ισχύ, την παλιά της ισχύ στο άρθρο την παλιά του ισχύ στο άρθρο 42 θα πρέπει να δούμε ποια είναι η, η γενική αρχιτεκτονική του, δικαιο, του δικαίου και ίσως να τροποποιήσουμε τον κανονισμό 1184 του 2006, γιατί ο κανονισμός αυτός ε, δικαιολογούνταν το 1962, αλλά δεν δικαιολογείται πια. Κατά τη γνώμη μου, μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να οδηγήσει σε τροποποίηση και μια λήψη υπόψη της ιδιαιτερότητας ε, της γεωργίας. Ευχαριστώ. Grazie. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την ε, καθηγήτρια Ντελκόντ από το Πανεπιστήμιο της Νάντης. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα τα όσα ακούσαμε. Ε, ιδιαίτερα ο εισηγητής μας, ο Μισελ Ταντάν, ε, για την ενιακό ε, άκουσε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και καλό είναι να ακούσουμε και τη φωνή των καθηγητών που υποστηρίζουν το έργο μας. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα τα όσα ακούσαμε, χρήσιμα και διευκρινίζουν και πάρα πολλές πτυχές. Ευχαριστώ βέβαια και τους υπολείπους που συμμετέχουν σε αυτό το σημαντικό εργαστήριο. Θα ξεκινήσει τώρα η συζήτηση και κατόπιν θα σας ξαναδώσω φυσικά το λόγο προκειμένου να απαντήσετε στις ερωτήσεις των βουλευτών μας. Να ξεκινήσουμε αμέσως με τον Μισελ Νταντάν. Μισελ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την ομάδα που εκπώνησε αυτή τη μελέτη που μας παρουσίασε η κυρία Ντερκόντ και πιστεύω ότι όντως το θέμα του δικαίου ανταγωνισμού και το θέμα των εξουσιών των, των οργανώσεων των παραγωγών είναι πολύ σημαντικό στα πλαίσια της κοινή γεωρικής πολιτικής. Επειδή υπάρχει οικονομική κρίση και έχουμε όλο και λιγότερα χρήματα για να διαχειριστούμε την αγορά, θα πρέπει να διαθετήσουμε τα διάφορα μέτρα που έχουμε για να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα κρατικά κονδύλια. Μετά από αυτά που ακούσαμε, θα ήθελα να πω ότι το ισχύον για τη Γεωργία δίκαιο είναι πολύ πιο περιοριστικό από ότι το γενικό δίκαιο ανταγωνισμού. Είχαμε πολλά παραδείγματα και μάλιστα αυτό το δόγμα στηρίζεται στην ε, πρωτοπόρα πολιτική της ΚΑΠ όπου είχε τιμές ανατολισμού που κατήφθηναν την αγορά και που στόχο είχαν μια αναδιοργάνωση της ε, ευρωπαϊκής γεωργίας, λαμβάνοντας υπόψη φυσικά το γεωργικό εισόδημα. Τώρα, εμείς αποφασίσαμε να περάσουμε από μια πολιτική ρυθμισμένων τιμών σε μια πολιτική των αγορών. Και αυτό είναι το νέο δόγμα που ισχύει εδώ και μια εικοσαετία. Είναι λογικό λοιπόν να τροποποιήσουμε και να προσαρμόσουμε το δίκαιο ανταγωνισμού μας, όχι ιδιαίτερα στη γεωργία, αλλά τουλάχιστον να έχει αντίστοιχα χαρακτηριστικά όταν ε, αυτά που ισχύουν και για τους άλλους, κανόν, για τους άλλους τομείς και για τις άλλες αγορές. Μία από τις ιδιαιτερότητες της γεωργίας είναι ότι εξαρτάται από τις ανάγκες των πελατών. Οπότε μία από τις ερωτήσεις που καλούμαστε να απαντήσουμε είναι από τη στιγμή που εγκαταλείψαμε μία κρατική πολιτική, κεντρική πολιτική ε, διαχείριση των αγορών θα επιτρέψουμε στις ιδιωτικές πρωτοβουλίες είτε των επαγγελματικών οργανώσεων είτε των παραγωγών να αντικαταστήσει αυτή την κεντρική κρατική πολιτική. Και να απαντήσουμε ναι στην ερώτηση θα πρέπει να δώσουμε τα μέσα στους γεωργούς ε, να έχουν διαπραγματευτική ισχύ απέναντι στους συνομιλητές τους. Και δεν είναι μόνο θέμα ε, συσπήρωσης των γεωργών. Το θέμα είναι από τη στιγμή που συσπηρωθούν και από τη στιγμή που οργανωθούν να έχουν αρκετές εξουσίες για να μπορέσουν να υπερασπίσουν και τα δικά τους συμφέροντα αλλά και να μην βλάψουν τα συμφέροντα των καταναλωτών. Γιατί αν δούμε τους διάφορους τομείς, τη ζάχαρη για παράδειγμα, είδαμε ότι μετά την μεταρρύθμιση του 2006 μειώθηκαν οι τιμές. Και τη διαφορά την εισέπραξε ο κλάδος, αλλά για τον καταναλωτή δεν είχε καμία διαφορά η κατάσταση, ούτε και για τον παραγωγό. Και οι παραγωγοί και οι καταναλωτές ήταν τα θύματα του συστήματος. Εμείς δεν θέλουμε να βλάψουμε ούτε τους παραγωγούς, τους γεωργούς, ούτε τους καταναλωτές. Και πιστεύω ότι είναι πολύ εύλογα τα σχόλια και οι συστάσεις που μας έκανε η ομάδα των ομαμαθών, όπω περιλαμβάνονται στη μελέτη που μας παρουσίασαν. Ευχαριστώ, Μισελ. Συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον Μάρτιν Χόισλινγκ και μετά την Ελίζα Γέγκλα. Νομίζω ότι το βασικό είναι ότι οι προτάσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο σημείο αυτό δεν επαρκούν καθόλου και θα πρέπει να βελτιωθεί η πρόταση και ότι για τον κλάδο αυτό χρειαζόμαστε ιδιαίτερο ιδιαίτερη νομοθεσία σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό. Αυτό το υποστηρίζω. Να σας πω ότι επειδή συζητήσαμε και για το πακέτο για τα γάλα σήμερα το πρωί, αυτό που με κάνει εντύπωση είναι η επιχειρηματολογία ότι οι γεωργοί δεν μπορούν να δεσμεύουν μεγαλύτερο ποσό, ποσοστό από 5,5% για παράδειγμα της παραγωγής. Αφετέρου, γιατί να περιορίζουμε τους παραγωγούς γεωργούς όταν, για παράδειγμα, τα γαλακτοκομεία έχουν τέτοιες συγκεντρώσεις. Γιατί να περιορίζεται έτσι η αγορά. Και το ίδιο ισχύει και για το εμπόριο, αν το δούμε και λίγο παραπέρα. Και ε, αντιληφθήκαμε ότι ουσιαστικά δεσμεύεται ε, ο γεωργός. Αυτό δεν είναι αυτό που επιθυμούμε, ο αποτροστόχος μας. Θέλουμε να δώσουμε ευκαιρίες στην γεωργία και ότι υπάρχουν απαγορεύσεις για τον καθορισμό τιμών, αυτό είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, γιατί τι νόημα έχει μία σύμβαση αν δεν μπορώ ως παραγωγός να ορίσω τις τιμές μου. Και αυτό ισχύει και για τις οργανώσεις που θέλουν να μπορούν να καταδείξουν ότι, για παράδειγμα, σημειώνουν ε, κάποια επιτυχία. τα κρατη στο πακέτο για το γάλα τελικά κατέληξαν στο ότι δήλωσαν εθελούσια συμμετοχή. Και αυτό θα πρέπει να είναι σαφές, ότι θα πρέπει να είναι εθελοντική η συμμετοχή. να έχουν κάποια μέρη του κλάδου τη δυνατότητα, μάλλον το να έχουν κάποια μέρη, μέλη μόνο, το δικαίωμα να κάνουν τέτοιες συμβάσεις δεν ε, θα αποφέρει αποτέλεσμα. Το σημαντικό είναι, και αυτό που αναρωτιόμαστε, και αυτό το απευθύνουμε και στον Επιτροπό Ανταγωνισμού, κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμφωνούσε στο σύνολο με μια τέτοια πρόταση. Γιατί έχω την εντύπωση ότι στην ε, Επιτροπή ε, το δίκαιο του ανταγωνισμού πάντα το βλέπουμε από την πλευρά και από το πρίσμα του καταναλωτή. Για να αγοράζει, για παράδειγμα, ευθύνα ο καταναλωτής. Δεν βάζουμε δηλαδή στον επίκεντρο, στο επίκεντρο τον παραγωγό. Και γι' αυτό υπάρχει μια ανισορροπία και μου προκάλεσε έκπληξη το γεγονός ότι οι αρχές ανταγωνισμού επέκριναν αυτό το μικρό τμήμα που έχουμε για το γάλα σε ό,τι αφορά τις επιδράσεις ε, στην ε, αγορά. Και νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να συζητηθούν στην Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Ευχαριστώ η Ελίζαμπετ Γέγκελ και μετά η κυρία Μαγκίνης. Ελίζαμπετ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα συμφωνήσω η συζήτηση σήμερα το πρωί κατέδειξε εκ νέου με σαφήνεια ότι αφενός είμαστε υπέρ της απελευθέρωσης, ε, έχουμε και απελευθέρωση της αγοράς σε πολλούς τομείς, αλλά πάντα όταν προκαλείται κάποιο πρόβλημα, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τη ζήτηση, ποιο είναι το πλαίσιο, ποιες είναι οι δυνατότητες που έχουμε στα πλαίσια της ε, απελευθέρωσης. Αν σωστά κατάλαβα, είπατε ότι το δίκαιο του ανταγωνισμού είναι υπερκείμενο σε σχέση με το δίκαιο για τη γεωργία. Ότι δεν ισχύουν οι παλιές αρχές. Επίσης είπατε ότι η γεωργοί πρέπει να είναι πραγματική φορή στα πλαίσια ε, του ανταγωνιστικού πλαισίου στο μέλλον. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε λοιπόν την κατάσταση αυτή το πακέτο για το γάλα και η όλη συζήτηση για το γάλα κατέδειξε ότι δεν θέλουμε τέτοια ετελούσια συμμετοχή και θέλουμε εμείς ε, να, ε, να διαμορφώσουμε την κατάσταση. δύο πράγματα νομίζω πρέπει να σκεφτούμε. Καταρχάς ότι θα πρέπει να καταρτήσουμε ένα κατάλογο καταχρηστικών πρακτικών και να ξεκαθαρίσουμε τι θεωρούμε εμείς εδώ στην Επιτροπή μας άδικο και κατά δεύτερον όταν ε, λέμε ότι θα πρέπει να είναι παράγοντες ε, οι αγρότες, θα πρέπει να το δικαίωμα να είναι παράγοντες που δρούν. Και το πακέτο για το γάλα δεν τους το εξασφαλίζει αυτό. Θα μπορούσαμε από πλευράς μας να δημιουργήσουμε, να απαιτήσουμε ένα νομικό πλαίσιο στο οποίο τα βασικά νομικά ζητήματα του συμβατικού δικαίου σε ό,τι αφορά τους όρους προμήθειας, διαμόρφωσης των επιχειρήσεων μεταξύ των, ε, των συναλλαγών των επιχειρήσεων, να οδηγήσει σε μια σαφή λύση πανευρωπαϊκή, την οποία θα πρέπει να μεταφέρει κάθε κρατός μέλος σε εθνική νομοθεσία. Σε ό,τι αφορά τώρα προστασία, την προστασία του καταναλωτή, καταφέραμε τα, να ρυθμίσουμε τα πράγματα έτσι, και σίγουρα δεν θέλουμε να κάνουμε βήματα προς τα πίσω, αλλά χρειάζονται αυτές οι δυνατότητες. Θα μπορούσαμε να δώσουμε την αρμοδιότητα να τα ορίσει αυτά η Επιτροπή Γεωργίας για όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλυσίδας των τροφίμων. Ευχαριστώ η Μάριαν Μαγκίνης και μετά ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τους εμπειρογνώμονες ε, για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Νομίζω ότι θα πρέπει να μελετήσουμε όλες τις παρατηρήσεις που έγιναν για τον ανταγωνισμό και για τον τρόπο που συνδέεται με τη γεωργία και συμφωνώ και με τα σχόλια του Μισελ Νταντά για τα θέματα που έθιξε. Μία γενική παρατήρηση αφορά και κάτι που ακούσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα το πρωί και μια συνεδρίαση που έκανα το μεσημέρι στην οποία προέδρευα ε, και αυτό που λέγαμε με την Ελίζα Μπεθιέγκλη για την ε, αλυσίδα των τροφίμων. Μεταρρυθμίζεται η ΚΟΑ αλλά και παραλλήλου υπάρχει και αυτή η κατάσταση η οποία είναι μη ρεαλιστική, όπου ενδιαφερόμενοι κάθονται και συζητούν επί του ζητήματος με την Κομισιόν, το Κοινοβούλιο δεν εμπλέκεται άμεσα, τον Ιούνιο θα υπάρξει έκθεση και στο τέλος του έτους, όταν θα ολοκληρωθεί το έργο μας, θα υπάρχει πολύ πιο ουσιαστικό έργο οι εμπειρογνώμονε που μα μίλησαν το μεσημέρι στη συνεδρίαση έχουν ετοιμάσει μια έκθεση για το τι συμβαίνει επί του ζητήματο στα κράτη-μέλη και είναι σαφέ ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν πρόβλημα με την αδικία, τι αθέμητε πρακτικέ και τι δυσκολίε για του παραγωγού. Κάποιοι προσπάθησαν την να ακολουθήσουν την προσέγγιση τη ήπια νομοθεσία, αλλά οι περισσότεροι πιστεύουν ότι χρειαζόμαστε πιο αυστηρή νομοθεσία και πιέζουν προ αυτή την κατεύθυνση. Είναι σαφέ ότι οι αρχέ του, ε, του ανταγωνισμού και τολμώ να πω και η Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Ανταγωνισμού και η ε, ο τομέας της λιανικής πώληση δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να συνεχίσουμε το έργο μας γνωρίζοντας ότι συμβαίνει και κάτι εκ παρελίλου σε άλλου φόρουμ και να λάβουμε υπόψη και το τι κάνουμε εμείς εδώ και να φροντίσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα ζυμαδίζουμε, θα πηγαίνουμε προς την ίδια κατεύθυνση και μπορούμε να επηρεάσουμε και αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και είμαι βέβαιη ότι ο Μισελ Μπαρνιέ, ο Επίτροπος Τσιόλος και ο τρίτος Επίτροπος που εμπλέκεται σε όλα αυτά, ο Επίτροπος Ταγιάννη, Καταλαβαίνω ότι έχουν καλή πρόθεση και είναι προετοιμασμένοι να αναλάβουν δράση επί του ζητήματος, αλλά πρέπει ακόμα να δω τι ρόλο μπορούμε να διαδραματίσουμε και εμείς όλα αυτά. Ευχαριστώ. Σωστά, ευχαριστώ. Ο κύριος Άγνιου και κατόπιν ε, ο Αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Τρεις ερωτήσεις για το πάνελ δύο αφορούν τη χώρα μου, τη ε, Μεγάλη Βρετανία και η τρίτη είναι γενικής φύσεως. Εξετάζουμε τον τομέα ζάχαρη στη Βρετανία και δύο είναι οι οργανώσεις που έχουν κυριαρχή θέση. Και η μία εκ των δύο είναι η μόνη οργάνωση που διαπραγματεύεται εκ μέρους των παραγωγών για την επεξεργασία της ζάχαρης. Η Βρετανική ζάχαρη έχει και το μονοπόλαιο για την κατεργασία, η British Sugar ε, έχει το μονοπέλιο για την κατεργασία. Επομένω, πρόκειται για δύο οργανισμού και μόνον. Και το αποτέλεσμα δεν φαίνεται να είναι σκανδαλώδε. Η ζάχαρη πωλείται στα ράφια των σούπερ μάρκετ και δεν συζητάει κανένα πόσο πρέπει να πληρώσουν για τη ζάχαρη. Μπορείτε να με διαβεβαιώσετε ότι, ότι αυτό το σενάριο δεν απειλείται από τη νέα νομοθεσία. Δεύτερον, ο όρος προεξάρχουσα δεν έχει ε, καθοριστεί. Τι σημαίνει 50% της αγοράς ε, είναι παραπάνω αυτό το ποσοστό. Μήπως αυτή η νομοθεσία θα επηρεάσει τον ανταγωνισμό στη Βρετανία, θα την παραγωνίσει και θα επιβάλλει τη δική του την νομοθεσία. Και τρίτον, πιστεύετε ότι η νομοθεσία θα έχει αντίστοιχε επιπτώσει σε κάθε κράτο μέλο παρά το γεγονό ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλε διαφορέ ε, και σε μεγέθη ε, αλλά και σε νομοθεσία σε κάθε κράτο μέλο. Ευχαριστώ, Άγνιου. Ο Ζωζεμποβέ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα του επιτελείου της Νάντης ε, για το έργο της γιατί πραγματικά είναι διαφωτιστική αυτή η μελέτη, γιατί τώρα μελετούμε τα κείμενα της ενιαίας κοινή οργάνωσης αγοράς και μας χρειάζονται τέτοιου είδους ε, διευκρινήσεις και διαφωτιστικές μελέτες. Είναι πραγματικά περίεργη η σημερινή κατάσταση, γιατί βλέπουμε αφενός επιθέσεις και τις καταδίκες ε, ε, με μια σκανδαλώδη κατάσταση που έγινε με τους παραγωγούς κάποιων λαχανικών. Επίσης έχουμε τα γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουμε μία οργάνωση ε, αγοράς που αντιβαίνει στην οικονομική αποτελεσματικότητα. Επίσης ε, καταγγείλαμε σε μία έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εγκρίθηκε στην Ολομέλεια ε, το γεγονός ότι η υπεραξία ε, ε, μεταφερόταν προς τις μεγάλες αλυσίδες διανομής και το 31% περάσαμε στο 20% μόνο για τους παραγωγούς και διαπιστώνουμε και το πρόβλημα που υπάρχει με τους κανόνες αναγωνισμού. Αν εξετάσουμε το πρώτο, το αρχικό κείμενο του 62, θα μπορούσαμε να ανατρέξουμε και στη συνθήκη της Ρώμης του 57 και αν δούμε αυτή τη λογική με οργανωμένες τιμές, καθορισμένες τιμές, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ένα αξιοπρεπές ιερικό εισόδημα στους γεωργούς αντίστοιχο με αυτών των άλλων ε, κατηγοριών ε, επαγγελματιών, τότε το κείμενο είχε ένα νόημα, αλλά όχι πια σήμερα. Γιατί έχουμε νέους πια οικονομικούς κανόνες που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τη δημοσιονομική κατάσταση ε, και δεν μπορούμε πια να είμαστε συμβατοί με τη συνθήκη της Ρώμης. Ο Μεσέλ Νταντά, ε, όπως μας είπε, ε, καλό θα είναι να συσπηρωθούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αντισταχθούμε στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό επιδιώκουμε τώρα και θέλουμε πραγματικά να σημειώσουμε πρόοδο, να προχωρήσουμε, ώστε να έχουμε μια συνεκτική πολιτική και μια δημοσιονομική πολιτική που θα παρακολουθεί την οικονομική πολιτική. Αλλιώς ε, θα, γίνουμε, θα βγούμε τα θύματα αυτής της κατάστασης που δεν θα ενισχύσει τους παραγούς ή τους καταναλωτές παρά μόνο τις μεγάλες αλυσίδες διανομής. Ευχαριστώ τον Ζωζέ ευχαριστώ όλα τα μέλη που έλαβαν το λόγο. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, να δώσω και πάλι το λόγο στους καθηγητές, κυρίως την κυρία Ντελκόντε, αν θέλει να απαντήσει στα όσα της ε, τέθησαν και να την ευχαριστήσω και εγώ για την εξαιρετική τους δουλειά και εσάς και το συνάδελφο Γεναρέλη. Εξαιρετική δουλειά, πραγματικά ευχαριστώ. Ναι, καταρχήν να δώσω κάποιες απαντήσεις πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Καταρχήν, ως προς το πώς δικαιολογείται ο, ο περιορισμός, η του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθε των οργανώσεων παραγωγών. Γιατί επιβάλλοντας ε, το άρθρο 120, δηλαδή απαγορεύοντας την κατοχή πόσες θέσης, δημιουργείται ένας ε, διπλός προβληματισμός. Πέραν της ε, αντίφασης με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού, έχουμε και την αντίφαση με τους στόχους που επιδιώκουμε. Το γεγονό ότι περιορίζεται το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε των γεωργών δεν οδηγεί κατά ανάγκη σε μια διαρθρωτική συγκέντρωση των εκμεταλλεύσεων και άρα σε ένα κίνημα, σε μια κατάσταση που αντιβαίνει στην πολιτική της ανάπτυξης υπαίθρου που έχει στόχο τη διαφύλαξη της πολυμορφίας και του πλουραλισμού των εκμεταλλεύσεων. Είναι κάτι λοιπόν που μας κατέπληξε. Επιπλέον, ο έλεγχος των συγκεντρώσεων και ανάντη και κατάγγι ε, ουσιαστικά ευνοεί τις ε, μεγάλες ε, δομές, στους μεγάλους ομίλους που ήδη ε, έχουν ε, δεσπόζουσα θέση. Οπότε δημιουργούνται διάφορα παράδοξα εδώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη γεωργία και τον ανταγωνισμό. Το θέμα δεν είναι να πούμε ότι η γεωργία εκπίπτει του πεδίου εφαρμογή του ανταγωνισμού ή θα πρέπει ε, να επωφελείται από δικαιολόγητε εξαιρέσει ή να εξαιρείται από το δίκαιο του ανταγωνισμού. Αλλά έχουμε δυνατότητα οριζόντιας και κάθετης εισπύρωσης των παραγωγών. Και αυτό είναι ε, βασικό κανόνα του δικαίου ανταγωνισμού, να επιτρέψουμε και στους γεωργού να έχουν κάποια νόμιμα στη διάθεσή του και συνθήκες διαφάνειας προκειμένου να διαμορφωθεί μια ομοιόμορφη αγορά. Κάτι που είναι απαραίτητη προπόθεση για μια αγορά στην οποία θα ισχύει ο ανταγωνισμό. Δεν είναι αδικαιολόγητη η υπέρμετρη λοιπόν αυτή, ε, αυτή η απέτηση για κάποιες εξαιρέσεις. Και δεν ξεφεύγουμε και από την οικονομική λογική. Τελευταία παρατήρηση πριν δώσω το λόγο στου είναι ότι όταν λέμε ότι η γεωργία είναι οικονομικός κλάδος, αυτό ισχύει, αλλά πρόκειται για έναν οικονομικό κλάδο που επιτελεί και κοινωνική λειτουργία. Δεν είναι μόνο η παραγωγή και η ανταλλαγή κάποιων εμπορεύσιμων αγαθών. Παρόλο που δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο ρητά στη συνθήκη, η γεωργία επιτρέπει πάνω απ' όλα την υλοποίηση του δικαιώματος ε, της ε, διατροφής στον πολίτη. Οπότε έχει και κοινωνική λειτουργία, έχει και περιβαλλοντική λειτουργία και ε, ανάπτυξη, λειτουργία ανάπτυξη πέθρου. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε την γεωργία ως πετρέλαιο, κάτι που κάνει η, ο γαλλικός οργανισμός συγκρίνοντας τη γαλακτοκομική παραγωγή με την ε, παραγωγή πετρελαίου. Είναι αγαθά βέβαια τα προϊόντα τα γεωργικά, αλλά διαφορετικά από τα υπόλοιπα εμπορεύσιμα αγαθά, μια και περιέχουν και μια κοινωνική λειτουργία. Νομίζω ότι με βάση αυτή, αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Γεωργίας μπορούμε να εφαρμόσουμε και με ιδιαίτερο τρόπο σε αυτήν το δίκαιο ανταγωνισμό. Ευχαριστώ. Καθηγητά Γιαναρέλη. Ναι, θα ήθελα να απαντήσω για να κάνω μια διευκρίνηση γενικού χαρακτήρα στις ερωτήσεις που ετέθησαν από τον ε, την Αγγλίδα Ευρωβουλευτή, συγγνώμη, από τον κύριο Άγνιου, ιδίω για το παράδειγμα της ζάχαρης που μας έφυξε. Ε, το ερωτηματικό αυτό μας επιτρέπει να εξηγήσουμε ε, την έννοια της ε, επιχειρηματολογίας μας και τους περιορισμούς φυσικά της παρουσίας μας. Λαμβάνοντα υπόψη την πραγματικότητα του σημερινού βιομηχανοποιημένου κόσμου, ξεκινήσαμε από το σκεπτικό ότι η παραγωγή διαρθρωτικά είναι ε, οικονομικά ε, οικονομικοί φορείς πολύ πιο ασθενείς από τους άλλους ή λόγω της ιδιαιτερότητας των αγορών τους. Για πολλά χρόνια προσπαθούσαμε να προστατεύσουμε και να αντιδράσουμε σε αυτή την αδυναμία με πολιτικές τιμών. Ε, κατά κάποιο τρόπο δηλαδή προσπαθήσαμε να ε, λύσουμε τα προβλήματα της αποτυχίας των αγορών μέσω του ελέγχου των τιμών. Αυτή τη στιγμή κατέρευσε ο μηχανισμός του ελέγχου των τιμών. Ο μόνος τρόπος ε, που εντοπίστηκε για να προασπίσουμε τους γεωργούς είναι οι συνεταιρισμοί και επομένως δομές οι οποίες μπορούν να εξισορροπήσουν ε, την συμβατική εξουσία που ε, ασκούν στους εταίρους τους. Ε, η ανησυχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ είναι ότι παραδόξως ο, ο μηχανισμός αυτής της προεξάρχουσας της δεσπόδουσας θέσης στην αγορά δημιουργεί ένα στοιχείο ε, δυσμένειας ε, του γεωργικού τομέα σε σχέση με τους άλλους τομείς. Διότι στο άρθρο 102 της συνθήκης ε, στους κανόνες του ανταγωνισμού απαγορεύεται η κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης, αλλά δεν απαγορεύεται σε μια επιχείρηση ευρωπαϊκού επίπεδου να έχει δεσπόζουσα θέση και μπορεί να δημιουργηθεί μια κατάσταση ενώπιον της οποίας στη γεωργία δεν θα μπορεί κάποιος να έχει δεσπόζουσα θέση. Και επομένως η αντίρρηση της συναδέλφου είναι ότι θεωρητικά θα μπορούσαμε να ευνοήσουμε τη δημιουργία όχι στην αγορά, αλλά μιας εδαφικής δομής η οποία θα εναγκαλίζει τους γεωργούς, ουσιαστικά δηλαδή θα είμαστε αντίθετοι στην ε, πολιτική της υπαίθρου. Αυτό λοιπόν το οποίο θα πρέπει να μας ανοσυχεί είναι η κατάχρηση της δεσπόδουσας θέσης και είναι παράδοξο να προσπαθούμε να απαγορεύσουμε στην γεωργία τη δημιουργία ε, συνεταιρισμών παραγωγών. Το άλλο επιχείρημα είναι ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μην συγχαίουμε τους ε, ε, επιχειρησιακούς οργανισμούς ε, της της νομοθεσίας κατά της δημιουργίας trust με την ε, νομοθεσία που ε, έχουμε σε εθνικό επίπεδο. Στην ε, χώρα τους ο καθένας εκτός από την κοινοτική νομοθεσία είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει και την νομοθεσία στη χώρα του, ό,τι ισχύει. Το παράδειγμα που έκανε ο συνάδελφός σας για την British Sugar και τη συγκεκριμένη δράση της. Εάν υπήρχε μία δεσπόζουσα θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο με κατάχρηση, τότε θα βρισκόμασταν ενώπιον μιας υπόθεσης εφαρμογής ε, και παραβίασες του νόμου του ανταγωνισμού ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν όμως είμαστε απλώς ένα φαινόμενο το οποίο ουσιαστικά αφορά αποκλειστικώ και μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο, ισχύει απλώς και μόνο η νομοθεσία ανταγωνισμού του Ηνωμένου Βασιλείου. Επομένως, σε επίπεδο νομοθεσίας ανταγωνισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργείται μια αναμαλία. Ουσιαστικά ε, προβλέπουμε απαγόρευση αναγνώρισης συνεταιρισμών που έχουν ε, δεσπόδουσα ή κυρίαρχη θέση. Εδώ δημιουργούνται διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων και οργανώσεων παραγωγών που δεν είναι ε, οι ίδιοι αλλά εντός της ευρωπαϊκής νομοθεσίας θεωρούνται ίδιοι. Ξεκινάμε από το σκεπτικό λοιπόν ότι ο γεωργός ε, θα πρέπει να την χάνει ιδιαίτερης προσοχής και να έχει ε, και δικαίωμα ε, προώθησης για να προστατεύσουμε τους ίδιους τους γεωργούς και βρισκόμαστε ενώπιον μιας νομοθεσίας που συμπεριφέρεται στο γεωργικό κόσμο, κυρίως τους συνεταιρισμούς παραγωγών που είναι η μόνη απάντηση που έχουν οι γεωργοί, δεδομένου ότι ως προς τις τιμές δεν έχουν καμία δυνατότητα να δράσουν, να μην μπορούν ε, τελικώς να χρησιμοποιήσουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσαι και να αποκτήσουν δεσπόζουσα θέση. Η ένσταση λοιπόν θα μπορούσε να είναι ότι μια ισχυρή ε, οργάνωση παραγωγών θα μπορούσε να επηρεάσει ακόμα και τις τιμές σε τελικό επίπεδο. Αλλά αυτή η ένσταση δεν ισχύει, διότι τη σήμερα ημέρα βρισκόμαστε ενώπιον ενός γεωργικού τομέα αποδυναμωμένου και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των τιμών παραγωγής και των τελικών τιμών, διότι υπάρχουν οι ενδιάμεση, οι οποίοι είναι ολιγοπόλια και παρεμβαίνουν. Και εδώ είναι το σημείο στο οποίο κανονικά θα έπρεπε να παρέμβουμε. Επομένως, ο ισχυρό προστατευτισμός είναι ίσως ένα μέσο που σε οικονομικό επίπεδο αγορά θα μπορούσε να προασπίσει τον πρωτογενή τομέα ενώπιον της ε, συμβατικής εξουσίας που έχει ο βιομηχανικός κλάδος. Και από εκεί και πέρα επαφίεται στο συνολικό επίπεδο ελέγχου της όλης αλυσίδας τροφίμων να αποφύγει, να αποτελέσει αυτό ζημία για τον τελικό καταναλωτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον καθηγητή Γιαναρέλη, ευχαριστούμε και την καθηγήτρια Τελικών και όλη της την ομάδα. Ε, πραγματικά μας χαροποιεί ιδιαίτερα η συνεισφορά σας και αν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις Α, παρακαλώ, ζητώ συγγνώμη να δώσουμε τώρα το λόγο ε, στον κύριο Μπόντικελ για να ολοκληρώσουμε το πλαίσιο. Θα ήθελα να σχολιάσω αυτά που είπε η Γερμανίδα Ευρωβουλευτής για κάποιες συμβάσεις. Είπε ότι οι συμβάσεις θα πρέπει να επιβάλλονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. αναφερθήκαμε στις συζητήσεις που έγιναν για τις ενοχικές υποχρεώσεις. Η μοναδική νέα υποχρέωση στην πρόταση είναι το γεγονός ότι οι συμβάσεις είναι γραπτές, γιατί οι συμβάσει υπήρχαν και στο παρελθόν. Απλώ εμπίπτουν σε εθνικού κανόνες. Τώρα υπάρχει υποχρέωση και γραπτή σύμβασης. Επίσης, μα, μας προβλημάτισε η χρησιμότητα αυτών των συμβάσεων, ποιο θα είναι μάλλον το χρηστικό τους αποτέλεσμα και τι μπορούμε να συμπεριλάβουμε σε αυτές τις συμβάσεις. Ε, δεν υπάρχουν αλλαγές ό,τι αφορά τη φιλοσοφία της σύμβασης, μια και υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις ενημέρωσης και επίσης και κάποιες ένομες συνέπειες ε, έως και κυρώσεις όταν τηρούνται οι διατάξεις. Πάντως, θα μπορούσαμε να προβλέπουμε υποχρεωτική αναφορά πολλών πληροφοριών και πολλών θεμάτων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, αλλά αν δεν προβλέψουμε ταυτόχρονα και κυρώσεις, οι διατάξεις δεν θα έχουν ε, πρακτικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ωραία, ολοκληρώσαμε τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την εξαιρετική σας συνεισφορά. Νομίζω ότι σας αξίζει ένα χειροκρότημα. Adesso, colleghi, ehm, vi propongo... Τώρα, προτείνω να ε, κάνουμε τώρα το σημείο 15 στην ημερήσια διάταξη, την έκθεση της κυρίας Καλνιέτε, ε, σχόλια εκτός μικροφώνου, η Κομισιόν ε, μάλλον δεν ήθελε να λάβει το λόγο επί του ζητήματος. Έλεγα λοιπόν ότι θα κάνουμε το σημείο 15, θέσπιση του προγράμματος πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία Ορίζον 2020, συντάκτρια της νομοδότησης η κυρία Καρνιέτα, η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το επόμενο πλαίσιο για την έρευνα, που είναι γνωστό ως Ορίζον 2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ουσιαστική αύξηση του προϋπολογισμού για την έρευνα στο γεωργικό τομέα, ε, κυρίως στη βιοοικονομία. Η έρευνα και η καινοτομία είναι οι πιο σημαντικές από ποτέ αυτή τη στιγμή, διότι η πρόκληση είναι να παράγουμε περισσότερα, μολύνοντας, ρηπαίνοντας λιγότερο. Το λόγο έχει κυρία Καλνιέτε. Ε, καλωσορίζω και το εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σάντρα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πρόγραμμα αυτό συνοψίζει όλα τα αποτελέσματα στον τομέα της έρευνας και χωρίς αυτό δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε την καινοτομία στην Ευρώπη, δεν θα μπορέσουμε να προωθήσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το κεφάλαιο του προγράμματος Ορίζοντος 2020, το οποίο συζητάμε σήμερα, να επικεντρωθεί κυρίως στην βελτίωση της βιοπικιλότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της σχετικής ανταγωνιστικότητας. Τα μέσα στον ορίζοντα του 2020 προβλέπονται συνολικά για τις έρευνες στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπονται για την ασφάλεια των τροφίμων, ισορροπημένη γεωργία, έρευνα θαλάσσια, τεχνική έρευνα, δύο έρευνα. 7,4 εκατομμύρια προβλέπονται. Έχουν ήδη δηλαδή προκαθοριστεί αυτή οι πόροι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ε, γεωργία. Θα ήθελα να τονίσω επίσης ότι η πολυτομιακή προσέγγιση στην εφαρμογή όλων των προγραμμάτων έρευνας είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών κέντρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον φυσικά ε, επεξεργάζονται ίδιους και παρόμοιους τομεί. Αυτό θα ωφελήσει όλες τις πλευρές. Η ζήτηση σήμερα για τρόφιμα σε παγκόσμιο επίπεδο αυξάνεται και χρειαζόμαστε όλο και πιο πολλούς φυσικούς πόρους για την παραγωγή των τροφίμων. Άρα δεν μπορούμε να αποτεχτούμε «30% των τροφίμων που παράγονται στις αναπτυσσόμενες χώρες να πετιόνται. Και για να επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό, χρειαζόμαστε μια πολυσύνθετη προσέγγιση, μια πολυσύνθετη προσέγγιση η οποία θα βασίζεται στην έρευνα. Να σας ε, πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σκοπεύει να υποστηρίξει μια κοινωνικο-οικονομική μελέτη, όπου θα τονίσετε και ο βιολογικός παράγοντας. Είναι σημαντικό λοιπόν να βρεθούν μοντέλα, να υποστηριχθούν ε, ε, πρωτοβουλίες που θα έχουν ε, θετικό αντίκτυπο. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να τονίσω ότι πρόκειται να συνεργαστώ με τους σκιώδες εισηγητές και είμαι βέβαιη ότι τελικά όλοι θα καταρτήσουμε μια ισόρροπη γνωμοδότηση. η οποία τελικά θα ωφελήσει και την αρμόδια επί της ύλης Επιτροπή, την Επιτροπή Βιομηχανία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Αν υπομονώ να ακούσω και τα σχόλιά σας. Μάλιστα. Ας περάσουμε στη συζήτηση. Ευχαριστούμε την κυρία Καλνιέτε για την εισαγωγή που μας έκανε. η κυρία Ράιμερς παρακαλώ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ καταρχάς για την παρουσίαση αυτή της γνωμοδότησης και του προγραμματός πλαισίου. Εγώ έχω συναντηθεί με διάφορα πανεπιστήμια και αυτό που μου επισημάνθηκε είναι ότι είναι ενθουσιασμένη για την διεθνική συνεργασία, αλλά το πρόβλημα κάθε φορά είναι ε, το τεράστιο διοικητικό κόστος για κάθε πανεπιστήμιο. Και νομίζω ότι θα πρέπει να προσέξουμε όταν ε, συμμετέχουν πανεπιστήμια να απλοποιούμε τις διαδικασίες και το σχετικό διοικητικό έργο. Ξέρουμε ότι η έρευνα θα πρέπει να είναι δημιουργική. Η έρευνα σημαίνει άλλωστε το να αποδείται κανείς σε άγνωστους ε, τομείς. Θα πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν να μην είμαστε υπερβολικά αυσταίοι, να μην αποθαρρύνουμε την όλη έρευνα. Φυσικά θα πρέπει να υπάρχει κάποιος έλεγχος για τα κονδύλια που διαθέτουμε γιατί πρέπει να δικαιολογούμε όλα αυτά τα έξοδα. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν κάποιο πιο ευελικτό τρόπο. Για την γεωργία είναι σημαντικό να δούμε στο πρόγραμμα πλαίσιο ότι η έρευνα και η καινοτομία ε, έχουν να κάνουν και με τη μεταφορά της καινοτομίας. Πώς είναι δυνατόν να μεταφερθεί η έρευνα ε, η οποία έχει χρηματοδοτηθεί με ευρωπαϊκά κονδύλια, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί και στην πράξη και νομίζω ότι εδώ χρειαζόμαστε να προσεγγίσει η έρευνα, την πρακτική αν θέλετε χρησιμότητα, γιατί δεν είναι όλη η έρευνα, ξέρετε, εξίσου χρήσιμη για την πρακτική ε, εφαρμογή. Νομίζω ότι αυτό θα μας ωφελήσει ιδιαίτερα να αφιερώσουμε πιο πολλά κονδύλια για την έρευνα, γιατί ε, στο σημαντικά ε, έργα που έχουμε μπροστά μας στον τομέα της γεωργίας χρειαζόμαστε πιο πολλές πληροφορίες, μοντέρνες τεχνολογίες προκειμένου να καταφέρουμε με πιο λίγα μέσα να πετύχουμε πιο πολλά. Δεν θέλει άλλος κανείς το λόγο. Οπότε... Α, συγγνώμη, κυρία Μαγκίνα, στο μεταξύ ζήτησε το λόγο. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι Θέλουμε περισσότερα στοιχεία και καλύτερη γνώση της γεωργίας. Έχουμε γνώση, εμείς έχουμε συγκεντρώσει πολλές πληροφορίες, αλλά τις ε, μεταφέρουμε στους γεωργούς. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε καλύτερη ε, μετάδοση αυτών των πληροφοριών και των μελετών που γίνονται προς τους γεωργούς μας. Γνωρίζω ότι τα πανεπιστήμια είναι συναρπασμένα με αυτή την προοπτική ε, κονδυλίων Καλό θα ήταν λοιπόν να υπάρχουν προπολογισμοί και να γίνονται έρευνε, αλλά να έχουμε και συγκεκριμένο στόχο για τι έρευνε αυτέ, συγκεκριμένη εστίαση. Νομίζω ότι από αυτήν την άποψη χρειαζόμαστε κάποιε περαιτέρω γνώσει. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Ρανς Γκαρσία. Ευχαριστώ και χαίρομαι που λαμβάνω το λόγο αμέσω μετά την κυρία Μαγκίνες γιατί πραγματικά έχει απόλυτο δίκιο ελοχεύει ένας πολύ σημαντικός κίνδυνος ε, να πελαγοδρομήσουμε μέσα στην πληθώρα των γνώσεων και των πληροφοριών και να μην καταφέρουμε να τις ε, μεταβιβάσουμε στους γεωργούς, ε, στους παραγωγούς, στη βιομηχανία. Γιατί αυτό το πρόγραμμα για τον ορίζοντα 2020 προβλέπει δυνατότητα μετάβαση, μεταβίβασης των πληροφοριών και της γνώσης στην αγροεπισητιστική βιομηχανία. Οπότε ε, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την απειλή των διεθνών ε, συμφωνιών και τις κοινοτικέ προτιμήσεις που δίνουμε σε τρίτες χώρες είναι να ε, λάβει όλη αυτή την πολύτιμη γνώση που διαθέτουμε. Η μεταφορά λοιπόν της γνώσης, η μεταβίβαση της γνώσης θα πρέπει να εξασφαλιστεί από την έρευνα στους παραγωγούς, στον κλάδο. Επίσης, ό,τι πρόοδο έχουμε στην αγροεπισητιστική βιομηχανία, στις γεωγραφικές ενδείξεις, στις ονομασίες προέλευσης, στις, ε, ε, στα τοπικά προϊόντα. Ε, αυτές οι γνώσεις πρέπει να μεταφέρονται στους ενδιαφερόμενους, γιατί θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ποιότητα και στην πρωτοτυπία του ευρωπαϊκού προϊόντος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τώρα πραγματικά εξαντλήθηκε ο κατάλογος των αγορητών. Α, όχι. Πάλι. Συγγνώμη. Έχετε το λόγο. Συγγνώμη, δεν σας είδα προηγουμένως. Yes, thank you. Ναι, σας ευχαριστώ. Να υποστηρίξω αυτά που μόλις είπε η κυρία Μαγκίνες. Με ακούει, με ακίνει. Με ακούει. Γιατί με την υποστηρίζω εγώ. Ποιος εγώ. Υπάρχει κι άλλο ένα θέμα το οποίο τίθεται, ότι μπορεί κανείς να κάνει όλη την έρευνα που θέλει και μετά να δοκιμάσει τα αποτελέσματα και τελικά τα αποτελέσματα της έρευνας να τα καταργήσουν οι ακτιβιστές, οι πράσινοι, να τα καταστρέψουν. Αυτά συμβαίνουν συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Αρκετά αυστηρή κριτική του συναδέλφου, αλλά ο καθένα έχει το δικαίωμα τη γνώμη. του. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο τη Γενική Διεύθυνση Γεωργία. Παρακαλώ. Α, ε, Ο λόγο στον κύριο Χάλ, τον εκπρόσωπο τη Γενική Διεύθυνση Έρευνα. Ευχαριστώ, πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνετε τη δυνατότητα να πω δύο λόγια. Θα γνωρίζετε ήδη το γενικότερο πλαίσιο αυτό του νέου τομέα πρόκλησης, ο οποίος συμπεριλήφθη στο Horizon 2020, με αυξημένο προπολογισμό σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα πλαίσιο, ουσιαστικά έχει διπλασιαστεί το ποσό, γεγονός που καταδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει την ε, πολύ μεγάλη σημασία και την ολαιόν αυξανόμενη σημασία αυτού του τομέα. Για να απαντήσω τώρα στις παρατηρήσεις που έγιναν ε, προσφάτως και να προσπαθήσω να εξηγήσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνειδητοποιεί πλήρως ότι η ανάγκη να υπάρχουν κατάλληλοι μηχανισμοί προκειμένου τα ερευνητικά αποτελέσματα να φτάνουν στον τελικό χρήση. Είτε αυτός είναι ο Γεωργός, είτε είναι ε, οι υπηρεσίες ε, συμβουλών, είτε είναι αγροτικές βιομηχανίες ή μεγαλύτερες κλίμακες βιομηχανία πρέπει να λαμβάνουν όλο το αποτέλεσμα. Και αυτό το συνειδητοποιούμε σε μεγάλο βαθμό και επίσης το νέο πακέτο για την έρευνα είναι ένα πακέτο έρευνας και καινοτομία στην ουσία. Έχουμε συγκεράσει ε, την καινοτομία με την έρευνα και έχουμε δώσει στην καινοτομία πολύ μεγαλύτερη σημασία από ό,τι στο παρελθόν. Το έχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως αυτό και θα λάβουμε βήματα ώστε στο μέτρο του δυνατού θα φροντίσουμε να εφαρμόζονται και στην πράξη τα αποτελέσματα της έρευνας. Όλα αυτά βέβαια προϋποθέτουν να ακούσουμε και τι έχουν να μας πούν οι γεωργοί και οι οργανώσεις των γεωργών και η κοινότητα της υπαίθρου για να γνωρίσουμε ποια είναι τα συγκεκριμένα προβλήματα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ε, που δεν τους επιτρέπουν να εξελιχθούν περαιτέρω. Ίσως και η έρευνα θα πρέπει να ανταποκρίνεται περισσότερο και στις απαιτήσει και στα αιτήματα της κοινωνίας της υπαίθρου και των γεωργών ε, για να μας βοηθήσουν και να σχεδιάσουμε και τα θέματα που θα παρουσιάσουμε. Επίσης θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι έχουμε και κάποιες ευκαιρίες για περαιτέρω εξέλιξη οι οποίες δεν είναι βραχυπρόθεσμα προβλήματα, αλλά μακροπρόθεσμα προβλήματα. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει την ευθύνη να έχει και ένα πιο μακρόπνο ε, όρομα και να μην ε, περιορίζεται στα αυτά τα δύο-τρία χρόνια τα οποία μπορεί να ενδιαφέρουν ε, περισσότερο τους περισσότερους γεωργούς. Σαφώς και σκοπεύουμε να ασχοληθούμε με τα θέματα της ανταλλαγής πληροφοριών και της διαβίβασης των πληροφοριών ε, καταλήλως, ώστε να συμπεριληφθεί, ε, μάλλον συγγνώμη, μέσω της συμπερίληψης και του τελικού χρήστη στη διαδικασία. Ε, τα περισσότερα προγράμματα σε γενικές γραμμές αφορούν πολλούς τομείς ε, και περιλαμβάνουν και πολλούς τέρους. Και μία από τις ωραίες πτυχές της ε, έρευνας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι μπορούμε να έχουμε ένα αμάλγαμα πολλών ε, ε, αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων από όλη την Ευρώπη, γεγονός που μας επιτρέπει να λάβουμε υπόψη ένα πολύ ευρωτερό φάσμα θεμάτων. αν παράδειγμα κάποιος θέλει να βελτιώσει τη γονιμότητα του εδάφους, μπορεί να είναι πολύ διαφορετική η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε στην Ισπανία από ό,τι στην Πολωνία, αλλά υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά που θα θέλουν να τα γνωρίζουν όλοι. Το μοντέλο λοιπόν για τι δραστηριότητες τη κοινή έρευνας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσον αφορά τώρα τα σχόλια για την απλούστευση, ναι πράγματι αυτό είναι και ένα από τα ουσιαστικά στοιχεία αυτής της ε, δέσμης μέτρων. Η ε, Γκένκαν Κουίν ε, το έχει διευκρινίσει αυτό, θέλει να συμπεριληφθεί αυτό και στο ε, νέο ε, πακέτο και θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι τμήμα της διαδικασίας. Και όλα αυτά εντάσσονται στην Δέσμη μέτρων και πολλά μέτρα εξετάζονται σε μια απόπερα απλούστευσης αυτής της περίπλοκης ε, διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την οποία επικριθήκαμε πολύ στο παρελθόν. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι προκειμένου να υπάρχει αυτή η στενότερη σχέση με την κοινότητα της Υπέθρου και τους γεωργούς, ε, συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τους συναδέλφους από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και ιδίω σε αυτό το πλαίσιο της προτονόμενης αυτής ε, σύμπραξης ε, έρευνας και καινοτομίας. Και εδώ ε, θεωρούμε ότι υπάρχει περιθώριο να αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ των κονδυλίων και των ταμείων για τη γεωργία και του ορίζοντα 2020 και τα, τα κονδύλια για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Και εδώ περιμένουμε να έχουμε και σημαντικά ωφέλη από αυτή την τόσο στενή συνεργασία που έχουμε με τους συναδέλφους από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας οι δραστηριότητες του προγράμματος θα είναι, αποτελούν αντικείμενο συνδιαχείρισης μεταξύ των δύο γενικών διευθύνσεων, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και αυτή τη στενή σχέση που σας ανέφερα μεταξύ της ανάπτυξης υπαίθρου και των γεωργών. Θα σταθώ σε αυτά κύριε Πρόεδρε. Εάν υπάρχουν και άλλα συγκεκριμένα ερωτήματα θα προσπαθήσουμε να τα απαντήσουμε είτε εγώ από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνα και Καινοτομίας είτε οι συνάδελφοι από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς να υποβάλει ερωτήσεις ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον εκπρόσωπο είτε της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας είτε της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας. Δεν βλέπω κανέναν, οπότε να ξαναδώσω το λόγο στην εισηγητριά μας. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλές ερωτήσεις θα είχα. Θα ήθελα σε κάθε περίπτωση να ευχαριστήσω τους συναδέλφους γιατί εξέφρασαν τις αμφιβολίες που είχα και εγώ κατά την πρώτη ανάγνωση του εγγράφου. Να ευχαριστήσω επίσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το γεγονός ότι συνειδητοποιεί ότι υπάρχουν τα προβλήματα αυτά και για το ότι αναζητά τις καλύτερες λύσεις. Το μόνο που απομένει είναι πραγματικά να ελπίσουμε ότι θα συμβεί αυτό. Το ελπίζω άλλωστε, ε, το εύχομαι και σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές μας εργασίες και κατά τη σύνταξη της έκθεσης και την ψηφοφορία της, την ψήφιση της έκθεσης αυτής. Ελπίζω ο Horizon 2020 να σημαίνει και να φέρει τέτοιες προτάσεις για τους γεωργούς που θα οδηγήσουν στην καλύτερη δυνατή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερής της διάταξης. Δεν ξέρω αν έχει καταφθάσει ο προσκεκλημένος μας τον ε, καλωσορίζω θερμότατα τον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον κύριο Κρέτα, για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις προτάσεις μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής. Λίγα λεπτάκια για να ετοιμαστείτε, κύριε Κρέτα. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ε, merci. Ε. Σας ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση προκειμένου να σας παρουσιάσω την ε, γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που αφορούν τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Η γνωμοδότηση αυτή αφορά τα τέσσερα βασικά σχέδια κανονισμού που χαρακτηρίζουν την ε, μεταρρύθμιση αυτή. Αυτές οι προτάσεις κανονισμού περιλαμβάνονται και στην ετήσια έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου αλλά και στις ειδικές εκθέσεις ε, για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Σήμερα θα περιορίσω την παρουσίασή μου σε τέσσερις ε, άξονες. Σε τέσσερα βασικά σημεία. Το πρώτο σημείο αφορά την απλούστευση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ως προς το σημείο αυτό θα ήθελα να παρατηρήσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να λάβει υπόψη κάποιες παρατηρήσεις του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και του Ελεκτικού Συνεδρίου για την απλοποίηση. Και θα σας δώσω δύο παραδείγματα αυτής της προσπάθειας ικανοποίηση ικανοποίησης του αιτήματο απλούστευσης. Καταρχήν ε, θεσπίστηκε το καθεστώς των βασικών πληρωμών που αντικαθιστά με ένα νέο σύστημα δύο προηγούμενα διαφορετικά συστήματα. Το, το καθεστώς ενιαίας πληρωμής και το καθεστώς πληρωμής με βάση την επιφάνεια που ίσχυε στις περισσότερες χώρες, στις χώρες που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2004. Το 2004. Πρόκειται λοιπόν για μια απλούστευση, μια και ένα καθεστώς αντικαθιστά δύο προηγούμενα. Άλλωστε το καθεστώς του, των ενιαίων πληρωμών έλαμβανε ε, ε, τη μορφή 20 διαφορετικών τύπων και τώρα πια αντικαθίσταται από ένα ενιαίο καθεστώς ε, βασικής πληρωμής. Αναφυσβήτητη λοιπόν πρόοδος ως προς το στόχο της απλούστευσης. Δεύτερη πρόταση, απλοποιημένο καθεστώς για τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Για τα υπόλοιπα σημεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε το πρόβλημα και πρότεινε πρότεινε μεν κάποιες λύσεις που κατά τη γνώμη του ελεκτικού συνεδρίου θα είναι δυσεφάρμοστες στην πράξη. Και εντός λίγο θα σας δώσω και κάποια παραδείγματα για να τεκμηριώσω αυτή την άποψη. Πάντως, γενικώ το ελεγκτικό συνέδριο θεωρεί ότι οι νέες νομοθετικές διατάξεις της ΚΑΠ εξακολουθούν να είναι περίπλοκες. Και θα σας αναφέρω τρία παραδείγματα για να σας εξηγήσω τι εννοώ. Πρώτο παράδειγμα αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου. Το προτινόμενο πλαίσιο διατηρεί τα έξι επίπεδα κανόνων που πλαισιώνουν αυτές τις δραστηριότητες που υπήρχαν και προηγουμένως. Υπήρχαν στο παρελθόν από το Γενικό Κανονισμό για τα Διαρθρωτικά Ταμεία μέχρι τις Εθνικές Νομοθετικές Διατάξεις που συγκεκριμενοποιούν τις, α, τους όρους εφαρμογής των μέτρων ανάπτυξης της υπαίθρου. Δεύτερο παράδειγμα, ερεσιμότητα. Το ελεγκτικό συνέδριο θεωρεί ότι η αναδιαργάνωση του κανονιστικού πλαισίου, του νομοθετικού πλαισίου της πολιτικής αιρεσιμότητας, ναι μεν ε, περιλαμβάνει μια απλούστευση, γιατί μειώθηκε ο αριθμός των διατάξεων, η απλούστευση όμως αυτή είναι μόνο φαινομενική, γιατί στην ουσία ε, δεν υπάρχει ουσιαστική, δεν υπάρχει πραγματική απλούστευση. Τώρα, το θέμα των ενεργών γεωργών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να εστιάσει καλύτερα τις ενισχύσεις προς τους γνήσους, τους ε, πραγματικούς, αυθεντικούς γεωργούς, ε, τους ενεργούς γεωργούς όπως τους χαρακτηρίζει. Και από αυτή την άποψη συμφωνούμε με την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπής να γίνει καλύτερη στόχευση των ενισχύσεων προς τους ε, γεωργούς που είναι πραγματικά γεωργοί, που ασχολούνται πραγματικά με τη γεωργία. Αμφιβάλλουμε όμως αν το κατά πόσο τα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον κανονισμό μπορούν να εφαρμοστούν και εμπράκτος και μάλιστα με αποτελεσματικό τρόπο η εκτίμηση του ηλεκτρικού συνεδρίου είναι ότι ίσως ο κανονισμός ε, δώσει ένα γενικό ορισμό για το τι εστί ενεργός γεωργός και να αναθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την συγκεκριμένη διαχείριση αυτής της νομοθεσίας προκειμένου να την προσαρμόσει στην ε, πολυπλοκότητα και την πολυμορφία των ε, περιπτώσεων που διαπιστώνουμε στην πράξη. Κατά τη γνώμη του Ελεκτικού Συνεδρίου είναι αδύνατο να καλύψουμε σε έναν ορισμό όλες τις ε, συγκεκριμένες εκφάσεις της γεωρικής δραστηριότητας και μάλιστα σε ένα γενικό νομοθετικό κείμενο. Ο δεύτερος άξονας της παρουσίασής μου, δεύτερο σημείο, είναι οι στόχοι της κοινή γεωργικής πολιτικής. Θεωρούμε ότι οι νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν δίνουν μια ξεκάθαρη απάντηση ως προς τη συμβολή της ΚΑΠ, δηλαδή τι θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε με τις δαπάνες της κοινή γεωργικής πολιτικής. Δεν δίνεται μια ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, εξακολουθούν να βασίζονται, όπως και στο παρελθόν, στα στο ύψος των διαφόρων κονδυλίων και στους όρους χορήγησης των κονδυλίων και δεν ε, αναφέρουν ούτε τα αποτελέσματα που επιδιώκονται, ούτε το πώς θα καταμετρηθούν. Και η μετάβαση από μια πολιτική μέσων σε μια πολιτική αποτελεσμάτων ήταν και η αρχική υπόσχεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το έτοιμο που είχε λάβει από τα διάφορα θεσμικά όργανα πιστεύουμε ότι αυτή η αλλαγή προσανατολισμού που είχε θεωρητικά αναγγελθεί δεν έχει ένα πρακτικό αντίκρισμα στις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και θα σας αναφέρω εδώ τέσσερα παραδείγματα για τον καθορισμό των πραγματικών στόχων της κοινή γεωργικής πολιτικής, σε ό,τι αφορά τις άμεσες πληρωμές, για παράδειγμα. Το ελεγκτικό συνέδριο θεωρεί ότι δεν αναφέρεται τίποτα ως προς τους στόχους που εξυπηρετούν οι άμεσες πληρωμές στο διατακτικό του κανονισμού. Όχι μόνο δεν αναφέρεται τίποτα ως προς τους στόχους των άμεσων πληρωμών, αλλά δεν αναφέρεται τίποτα και ως προς τα αποτελέσματα που περιμένουμε από τις άμεσες πληρωμές. Ενώ περιμέναμε να γίνεται μια αναγγελία και μια συγκεκριμενοποίηση των στόχων. Δεύτερο παράδειγμα. Η κατανομή της ενίσχυσης μεταξύ των δικαιούχων. Ούτε και εδώ αναφέρεται κάποιο συγκεκριμένο στόχος. Η κατανομή των ενισχύσεων στηρίζεται, όπως και σήμερα, σε μεγάλο βαθμό στην ε, καλλιεργήσιμη επιφάνεια. Στις γεωργικές εκτάσεις δηλαδή. Ναι, δεν προτείνονται κάποιες μικρές αλλαγές, για παράδειγμα, διευκρινίζεται ότι οι γεωργοί των μειονεκτικών περιοχών και οι νέοι γεωργοί θα τύχουν ε, μια συμπληρωματική ενίσχυση ένα εκτάριο. Αυτό ίσω είναι ένα έμεσο τρόπο για να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη διάζουσα κατάσταση ορισμένων ε, γεωργών. Παρ' όλα αυτά, παρά, παρά, παρά αυτά τα δύο παραδείγματα που είναι θετικά κατά τη γνώμη μου, το ελεγκτικό συνέδριο κρίνει ότι το καθεστώς ε, χαρακτηρίζεται από μια εσωτερική αντίφαση που προϋπήρχε στο καθεστώς των, της ενιαίας πληρωμής. Δηλαδή, αφενός θέλουμε να στηρίξουμε το ατομικό εισόδημα των γεωργών, αφετέρου όμως δεν προσαρμόζουμε αυτή την ε, στήριξη στην ιδιαιάζουσα κατάσταση των εκμεταλλεύσεων. Ούτε λαμβάνουμε υπόψη την πολυμορφία των δαπανών που έχουν ε, να αναλάβουν οι γεωργοί που παράγουν τα δημόσια αγαθά που περιμένουμε από αυτούς. Γιατί η παραγωγή τέτοιων δημόσιων αγαθών ε, ίσως έχει διαφορετικό κόστος ανάλογα με τη γεωγραφική ζώνη, τη χώρα που βρίσκεται μια γεωργική εκμετάλλευση. Δεν υπάρχει όμως ε, τέτοια διαφοροποίηση στις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, διαφοροποίηση των ενισχύσεων ανάλογα με το κόστος ε, παραγωγής αυτών των δημόσιων αγαθών που είναι τα γεωργικά προϊόντα. Τρίτο παράδειγμα. Αφορά την αιρεσιμότητα και την οικολογική συνιστόσα που προβλέπει ο κανονισμός οι στόχοι και τα αποτελέσματα της αιρεσιμότητας και του, της οικολογικής συνιστώσας των άμεσων πληρωμών δεν προσδιορίζονται με σωστό τρόπο. Δηλαδή, γνωρίζουμε αφενός ότι υπάρχουν κάποιες επιστημονικές μελέτες που καταδεικνύουν την ανάγκη και επισημαίνουν την αποτελεσματικότητα της, του προσδιορισμού των ζωνών οικολογικού ενδιαφέροντος. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τέτοιες ζώνες οικολογικού ενδιαφέροντος ή οικολογικής εστίασης. Για τη βιοπικιλότητα υπάρχουν πολλές μελέτες που συνηγορούν με τη χρησιμότητά της. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι στον κανονισμό. Ούτε προσδιορίζεται η επίπτωση της εφαρμογής αυτών των μέτρων τελευταίο παράδειγμα για τους στόχους αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου. Το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάπτυξη της υπαίθρου α, περιλαμβάνει μια σειρά στόχων και προτεραιοτήτων που είναι ποικίλη και πολύμορφη. Το ελεκτικό συνέδριο θεωρεί ότι η πολιτική ανάπτυξη υπαίθρου θα πρέπει να στοχεύει σε πολύ πιο απλούς στόχους και να είναι καλύτερα εστιασμένη αυτή η πολιτική. Έρχομαι τώρα στον τρίτο άξονα της παρουσίασης. Αφορά την ε, επιτήρηση του συστήματος εφαρμογής και ελέγχου των γεωρικών δαπανών στα κράτη-μέλη επιτήρηση που εξασφαλίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα κράτη-μέλη έχουμε δύο είδη οργανισμών που διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Πρόκειται για τους οργανισμούς πληρωμών αφενός και τους οργανισμούς ε, πιστοποίησης αφετέρου. Σε ό,τι αφορά τους οργανισμούς πληρωμής, έχουν εξουσιοδότηση, ειδική εξουσιοδότηση από τα κράτη-μέλη. Το ελεκτικό συνέδριο θεωρεί ότι επειδή σε τελευταίο βαθμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρμόδια για την εκτέλεση του προπολογισμού, θα πρέπει να μπορεί να επιβλέπει την εφαρμογή αυτών των οργανισμών ήδη από την αρχή τους, χωρίς να περιμένει να εντοπιστούν κάποιες ελλείψεις ή ατασταλίες. Θα πρέπει να ελέγχει λοιπόν, να επιβλέπει την εφαρμογή αυτών των οργανισμών, καθώς και την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων που χρησιμοποιούν αυτοί οι οργανισμοί. Σε ό,τι αφορά τώρα τους οργανισμούς πιστοποίησης, αυτοί δεν ε, λαμβάνουν εξουσιοδότηση από τα κράτη-μέλη, απλώς ε, γίνεται ορισμός ε, από τα κράτη-μέλη και εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί το έργο αυτών των οργανισμών για να βεβαιωθεί για την χρηστή διαχείριση των γεωργικών κονδυλίων θεωρούμε ότι και εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ακριβώνει το ρόλο των συστημάτων και τις επιδόσεις των οργανισμών πιστοποίησης. Σε ό,τι αφορά αυτούς τους οργανισμούς πιστοποίησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει επέκταση του ρόλου τους πέραν της αξιοπιστίας των λογαριασμών γιατί σήμερα οι οργανισμοί πιστοποιήσεων πιστοποιούν τους λογαριασμούς των οργανισμών πληρωμής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια επέκταση αυτού του ρόλου, προκειμένου να καλύπτει και την πιστοποίηση της νομιμότητας και του νομότυπου των πληρωμών. Κάτι που δεν ίσχυε μέχρι σήμερα. Το ελεκτικό συνέδριο θεωρείται κάτι τέτοιο αποτελεί μια χρήσιμη ενίσχυση του ρόλου και του έργου των οργανισμών πιστοποίησης αλλά μας εκπλήσει ο τρόπος με τον οποίο ε, μεταφράζει στο σχέδιο κανονισμού το στόχο της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σχέδιο κανονισμού προβλέπει ότι στο μέλλον οι οργανισμοί πιστοποίησης θα εκφέρουν ε, γνώμη όχι ως προς τους λογαριασμούς ε, των οργανισμών πληρωμής αλλά ως προς τη δήλωση αξιοπιστίας διαχείρισης του διευθυντού ουσιαστικά του οργανισμού πληρωμής. Εμείς επιμένουμε στη μεγάλη διαφορά που υπάρχει μεταξύ πιστοποίησης των λογαριασμών και πιστοποίησης της νομοτυπίας του νομότυπου και της νομιμότητας των λογαριασμών και ε, γνώμης ως προς τη δήλωση αξιοπιστίας που υπογράφει ουσιαστικά ο διευθυντής του οργανισμού πληρωμής. Νομίζω ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω. Τέταρτος άξονας, τέταρτο σημείο, ίσως χρειαστεί να μακρηγορήσω εδώ, αλλά σας διαβεβαιώ ότι είναι το τελευταίο σημείο. Καλύπτει δύο θέματα. Θέμα της εκαθάρισης των λογαριασμών και της... την περίπτωση όπου δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ε, για την ε, πληρωμή μιας ενίσχυσης. Σε ό,τι αφορά την εκαθάριση των λογαριασμών, το ελεκτικό συνεδρίο θεωρεί ότι ε, στόχος της διαδικασίας εκαθάρισης λογαριασμών απομακρύνεται από το στόχο και τον ορισμό το, της διαδικασίας αυτής όπως προβλέπει ο δημοσιονομικός κανονισμός και τα εκτελεστικά μέτρα του. Ο δημοσιονομικός κανονισμός, το άρθρο 53 αναφέρει το σημείο αυτό και ε, το άρθρο 42 ε, του εκτελεστικού κανονισμού. Αυτά τα δύο άρθρα θα έπρεπε να εφαρμόζονται κανονικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ελεκτικό συνέδριο λοιπόν υπενθυμίζει ότι ο γενικό στόχο τη εκαθάριση λογαριασμών είναι να επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει την τελική της ευθύνη σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού. Και ιδιαίτερα στην περίπτωση των γεωργικών δαπάνων, γιατί οι γεωργικές δαπάνες εκτελούνται με βάση το καθεστώς της κοινή διαχείρισης. Οπότε θα πρέπει να αναλάβει την ε, ευθύνη των δαπανών που γίνονται από οργανισμούς πληρωμής όμως, που είναι εθνικοί οργανισμοί. Αυτό και έχουμε τη διαδικασία της εκαθάρισης των λογαριασμών. Αυτή η διαδικασία σημαίνει ουσιαστικά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφενός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ορίσει το ε, ύψος των δαπανών που έγιναν νομότυπα και άρα θα επιβαρύνουν τον κοινοτικό προπολογισμό και αφετέρου, αντίστροφα, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απορρίψει τις δαπάνες που δεν συνάδουν με τους κανόνες. Αυτός ο καθορισμός όμως ε, του ύψους των δαπανών που θεωρούν νόμιμες και νομότυπες και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεωρήσει ότι μπορούν να επιβαρύνουν το κοινοτικό προπολογισμό. Ο καθορισμός αυτού του ποσού που είναι αιτήσιος, των αποδεκτών δηλαδή τακτικών δαπανών, δεν περιλαμβάνεται στον κανονισμό ως υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάτι που χρήζει διευκρίνηση κατά τη γνώμη του ελεκτικού συνεδρίου. Και πάλι στο θέμα τη εκαθάριση των λογαριασμών. Θεωρούμε, θεωρεί το ελεκτικό συνέδριο, ότι καμία από τι προτινόμενε τροποποίησει δεν πρόκειται να μειώσει την προσφυγή στις δημοσιονομικές διορθώσεις που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διορθώσει τους λογαριασμούς και να κάνει την εκαθάριση. Αυτή η παρατηρήση είναι πολύ σημαντική, γιατί το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει μία διαφορά μεταξύ δύο τομέων των κοινοτικών πολιτικών, των ενωσιακών πολιτικών. Σε ό,τι αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία, δηλαδή το ΦΕΝΤΕΡ, αυτά είναι τα γαλλικά ακρονίμια, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής. Σε ό,τι αφορά τον κανονισμό που καλύπτει αυτά τα διαρθρωτικά ταμεία, αυτός ο, ειδικός, αυτός ο κανονισμός προβλέπει ότι στο μέτρο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια καταποκοπή δημοσιονομική διόρθωση, τα κράτη-μέλη δίνονται να αποδείξουν ότι το ύψος της ατασταλίας που διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κατώτερο, είναι χαμηλότερο από την αξιολόγηση, την αποτίμηση που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορούν τα κρατημένα να ισχυριστούν ότι η καταποκοπή διόρθωση είναι υπερβολική και φυσικά θα πρέπει να τεκμηριώσουν αυτό τον ισχυρισμό τους. Αυτή όμως η επιλογή της αφισβήτησης της καταποκοπή διόρθωσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ισχύει για τη γεωργία και δεν καταλαβαίνουμε γιατί υπάρχει αυτή η διαφορετική μεταχείριση της γεωργίας. Τέλος, τελευταίο σημείο κάποιες παρατηρήσεις για, τις, για τη μείωση των ενισχύσεων. Τι θα πει μείωση των ενισχύσεων. Η μείωση που θα εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά υπολογισμό του θεωρητικού ύψους της ενίσχυσης, γιατί δεν συνέτρεξαν όλες οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση μιας ενίσχυσης ή επειδή ένας γεωργός ε, είχε αναλάβει υποχρεώσεις που δεν τήρησε ή δεν τήρησε ε, πλήρως για να ε, δικαιούται μία ενίσχυση στα πλαίσια της ε, ανάπτυξη υπαίθρου. Στην περίπτωση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάται να μειώσει το ύψο των ενισχύσεων. Θεωρούμε όμως ότι για το σημείο αυτό είναι πολύ συγκεχημένος ε, ο κανονισμός και μάλιστα το άρθρο 65 του κανονισμού είναι ιδιαίτερα σαφές και συγκεχημένο γιατί προτείνει ένα πολύ τεχνικό διαχωρισμό μεταξύ της μείωσης των πληρωμών αφενός και μιας κύρωσης ε, με τη μορφή μείωσης ε, πληρωμών αφετέρου. Πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε αυτό το διαχωρισμό και τι θα πει ακριβώς κύρωση. Δεν εξηγείται στον κανονισμό τι νόημα έχει αυτή η κύρωση. Βέβαια δίνεται μια εξήγηση λίγο παρακάτω στο άρθρο 97. Το άρθρο 97 μας λέει ότι οι κυρώσεις που έχουν τη μορφή μείωσης ε, πληρωμών δεν ε, έχουν ε, συνέπειες, δεν έχουν επιπτώσεις στην νομιμότητα της πληρωμής. Τι σημαίνει αυτό και αυτό το σημείο μας παραξενεύει, αν το έχουμε καταλάβει καλά. Σημαίνει ότι ένας δικαιούχος που παραβιάζει τις κανονιστικές διατάξεις θεωρείται παρόλα αυτά ότι δικαιούται το, ολόκληρη την πληρωμή. Αυτή η πληρωμή θεωρείται νομότυπη. Παρ' όλα αυτά, ο δικαιούχος θα κληθεί να επιστρέψει ένα τμήμα της ε, ενίσχυσης, ίσως και το σύνολό της, με βάση το μηχανισμό μείωσης, και επιπλέον ε, θα πληρώσει και κάποια πρόστιμα για παραβίαση του των κανόνων. Και αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Τι νόημα έχει το άρθρο 65. Τι νόημα έχει και το άρθρο 97. Χρειάζονται σημαντικές διευκρινήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα δύο αυτά σημεία. Οι μειώσεις των ενισχύσεων είναι σημαντικό ε, ζήτημα της ε, πολιτικής αιρεσιμότητας, γιατί μέσω της μείωσης πληρωμών εφαρμόζεται η αιρεσιμότητα. Εφόσον δεν τηρηθούν οι υποχρεώσεις της ε, και οι όροι της αιρεσιμότητας, δεν δικαιούστε πια το σύνολο της ενίσχυσης και άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει μια μείωση αυτής της ενίσχυσης. Αυτές οι μειώσεις όμως ε, αυτό που θέλω να τονίσω τουλάχιστον το ελεκτικό συνέδριο είναι ότι αυτές οι μειώσεις για αθέτηση των υποχρεώσεων, της των υποχρεώσεων που απορρέουν από την αιρεσιμότητα ή μάλλον διορθώνει ο μιλητής οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την αιρεσιμότητα είναι ένομες υποχρεώσεις όπως και οι υπόλοιπε που ε, ισχύουν για όλους τους γεωργούς προκειμένου να δικαιούνται το σύνολο της ενίσχυσης και θεωρούμε ότι η αθέτηση αυτών των υποχρεώσεων θα πρέπει να καθιστά παράνομη ή παράτυπη την καταβολή της πληρωμής, κάτι που δεν ισχύει, την καταβολή της ενίσχυσης. Δηλαδή υποχρεώσεις από την αρεσιμότητα, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την αρεσιμότητα, δεν θεωρούνται προϋπόθεση επιλεξιμότητας για να έχει κανείς πρόσβαση στις άμεσες πληρωμές. Και πάλι ω προ την αιρεσιμότητα. Το ελεκτικό συνέδριο διαπιστώνει ότι το σύστημα μείωση ενισχύσεω σε περίπτωση παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την αιρεσιμότητα αποδυναμώνεται από τι νέε διατάξει. Γιατί το γενικό ποσοστό μείωση, που είναι τουλάχιστον 30%, αυτό το γενικό ποσοστό μείωση δεν περιλαμβάνεται πια στο νέο σχέδιο κανονισμού. Θα σταματήσω εδώ λοιπόν τις λεπτομεριακές μου παρατηρήσεις θα ήθελα ε, εν κατακλείδη να σας υπενθυμίσω κάτι που γνωρίζετε, ότι η μεταρρύθμιση αυτή θα έχει και ένα διοικητικό κόστος, ιδιαίτερα για τα κράτη-μέλη. Για τα κράτη-μέλη είναι αυτά που διαχειρίζονται αυτούς, αυτές τις ταπάνες μέσω των οργανισμών πληρωμών και των οργανισμών πιστοποίησης, όπως είπα προηγουμένως, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη μελέτη επιπτώσεων προβλέπει ότι αυτό το διοικητικό κόστος ε, θα οδηγήσει σε μία αύξηση 15% της διαχείρισης των ε, μεσοπληρωμών. πληρωμών. Είναι αρκετά σημαντικό αυτό το ποσοστό της αύξησης. Και το Λεκτικό συνέδριο θεωρεί ότι δεν έχουν ε, δοθεί αρκετές πληροφορίες για να τεκμηριώνουν την ε, αντιστάθμιση αυτού του συμπληρωματικού κόστους από αντίστοιχη αύξηση της αποτελεσματικότητας ή της αποδοτικότητας. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Λυπούμε που μακρηγόρησα, αλλά πραγματικά είναι μεγάλο και το νομοθετικό και βρήκε το νομοθετικό πλαίσιο και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Κρετά. Ε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας, η γνωμοδότηση της, ε, ε, του ελεγκτικού συνεδρίου που να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από το ελεγκτικό συνέδριο. Από ό,τι ακούσατε είναι πολλά τα σημεία τα οποία έθεσε επιτάπητος ο κύριος Κρετά, ε, θέματα τα οποία πρέπει να πω κύριε Κρετάν ότι έχουν μεγάλη σχέση με τη συζήτηση που έχουμε εδώ εμείς στην Επιτροπή μας. Ε, πάν πολλές φορές έχουμε σταθεί στα σημεία αυτά από τον ενεργό γεωργό, από το κόστος ε, για την εφαρμογή του greening και για τα κρατη αλλά και για το πόσο πιο περίπλοκα γίνονται τα πράγματα για τους γεωργούς. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει εδώ ψωμί στη συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν μπορούμε να την ξεκινήσουμε αμέσω τη συζήτηση και στο τέλο ε, τη συζήτηση θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε στι ερωτήσει των συναδέλφων και φυσικά θα ακούσουμε και τι έχει να μα πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν το επιθυμεί. Ξεκινούμε από την κυρία ε, Κέστιγκερ και κατόπιν ε, η Μπρίτα Ρέιμερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ και εσά, κύριε Κρυτάν, για τι εκτιμήσει σα και κυρίω για τη δυνατότητα που μα δίνετε να διεξάγουμε τη συζήτηση αυτή μαζί σας, γιατί ασφαλώς είναι πάρα πολύ σημαντικές οι πληροφορίες αυτές, μιας και βρισκόμαστε στην διαδικασία συναπόφασης πλέον και έχουμε καθήκον να αμβλύνουμε πολλά από τα προβλήματα αυτά που αναφέρατε. Δυστυχώς ε, δεν συμμετέχουν σήμερα στη συνεδρίαση πολλοί συνάδελφοι, κυρίως όσοι συνάδελφοι θεωρούν ότι θα πρέπει να επιβάλλονται διαρκώ όλο και πιο πολλέ απαιτήσει ε, στην γεωργική πολιτική και νομίζω ότι αυτό στο παρελθόν έχει αποδειχτεί ε, επιζήμιο. Το συζητήσαμε και με τον Επίτροπο Τσιόλο στο θέμα αυτό της απλούστευσης της ΚΑΠ και μας λέτε και εσείς ότι το βασικό πρόβλημα είναι τα κράτη-μέλη. Ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει πολύ απλά πράγματα τα οποία τα κάνουν περίπλοκα στη συνέχεια τα κράτη-μέλη. Αυτό θεωρείται ότι ισχύει, γιατί ξέρω από το δικό μου κράτος ε, μέλος επικρατεί φόβος για εξωτερικές ε, παρεμβάσεις και γι' αυτό είναι πάρα πολύ αυστηρή η έλεγχη Μιλήσατε και για τις αρχές και τις υπηρεσίες επιστοποίησης από πλευρά σας. Υπάρχουν συγκεκριμένες λύσεις που έχετε να προτείνετε για την άμπληση των προβλημάτων αυτών. Συμφωνώ με την εκτίμησή σας σε ό,τι αφορά τα μέτρα για την οικολογική πράσινη συνιστόσα που προτάθηκε στην διάρκεια των μεταρρυθμίσεων θα πρέπει και η Γεωργία να πληρεί τις πολλαπλές αυτές, ε, τις πολλαπλούς αυτούς όρους ε, συμμόρφωσης. Αλλά μήπως κάνουμε τον απότερο σκοπό τελικά και συμφωνώ επίσης σε ό,τι αφορά τις ε, συμβάσεις εταιρική σχέσης. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να γίνει και πολύ πιο περίπλοκο το ζήτημα. Και είναι σαφές ότι και πάλι ε, υπάρχουν ατασταλείς και σε πολλές περιπτώσεις δεν εξαντλούνται οι πόροι. Ευχαριστώ. Η Μπρίτα και μετά Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που βρίσκεστε σήμερα εδώ στην Επιτροπή μας για να ε, παρουσιάσετε αυτή την έκθεσή σας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση για τις ε, βασικές πληρωμές και για το, την, την οικολογική συνιστόσα. Στην Επιτροπή Γεωργίας έχουμε ασκήσει έντονη κριτική στο θέμα αυτό γιατί δεν θέλουμε να ληφθεί μία απόφαση χωρίς να είναι σαφής η στοχοθέτηση. Τι θα λέγατε αν ήταν αυτή η οικολογική συνιστόση στο δεύτερο πυλώνα και αν υπήρχε ε, ε, συρρήκνωση στον πρώτο πυλώνα. Θεωρείτε ότι θα ήταν πιο εύκολο αυτό στην ε, ε, εφαρμογή. Πώς το εκτιμάτε σε ό,τι αφορά τους διάφορους στόχους στον τομέα της υπαίθρου. Μήπως λείπει το θάρρος ε, να παραδεχτούμε ότι χρειαζόμαστε μια καθαρά αγροτική πολιτική, χωρίς ε, πολιτική ε, κοινωνική, οικονομική. Να μην αποδυναμώνουμε δηλαδή τον ίδιο τον πυρήνα της γεωργικής πολιτικής για θέματα ελέγχου. Ξέρω τι φοβούνται οι γεωργοί και δικαίω εν μέρη, γιατί μια μικρή γεωργική εκμετάλλευση λειτουργεί διαφορετικά από ότι ένας μεγάλος όμιλος. Στην γεωργία μια εκμετάλλευση καλύπτει όλη την παραγωγή. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, μετά την τοπική υπηρεσία ελέγχου έχουμε και την ομοσπονδιακή, την εθνική, ενδεχομένως και η Ευρωπαϊκή Αρχή για να κάνουν ελέγχους. Και άρα από πλευράς ε, Γεωργού υπάρχει μεγάλη ανάγκη απλούστευσης. Άρα, να μην κοιτάμε μόνο τα συντήματα ελέγχου από πλευράς ε, διοικητικής, αλλά και από πλευράς του Γεωργού. Το ελεκτικό συνέδριο συμφωνεί ότι σε περίπτωση παραβιάσεων, είτε είναι οι θελημένες, ε, περιπτώσεις απάτης δηλαδή, που πρώτο, όντως πρόκειται για κατάχρηση των κονδυλίων. Ε, αλλά υπάρχουν και παραβιάσεις οι οποίες είναι περιστασιακές, είναι παρουσιάζονται σε περίπτωση που για παράδειγμα δεν λειτουργεί μια τεχνολογία. Υπάρχουν ε, και παράγοντες, ξέρετε, όπως ο καιρό που δεν επηρεάζονται από κανέναν και ευτυχώ ε, στη Γεωργία. Αυτά δεν προβλέπονται όλα στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέτοιε παραβιάσεις δεν μπορεί να οδηγούν απαραίτητο σε κυρώσει. Αυτό θα ήταν άδικο. Γιατί αυτό θα σημαίνει διπλή ε, τιμωρία του αγρότη και σε ό,τι αφορά την δραστηριότητά του και σε ό,τι αφορά τα κονδύλια που λαμβάνει. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση για αυτά. Ευχαριστούμε, Μπρίτα. Ρούμπιξ και μετά κύριε Μαγκίνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ, κύριε Κροτά, που έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε μαζί σας σήμερα. Συμφωνώ με πολλά από αυτά που αναφέρατε και η δική μου, ξέρετε, το δικό μου εκλογικό κοινό συμφωνεί γιατί εκπροσωπώ εδώ τη Λετωνία. Οι Λετωνοί λοιπόν, οι Γεωργοί, συχνά με ρωτούν το εξή. Και θέλουν σαφείς απαντήσεις. Αξιολογούν θετικά την ε, ενιαία διαμόρφωση των πληρωμών. Αλλά οι πληρωμές είναι πολύ διαφορετικές στο ύψος τους. Η γεωργοί στη Λετωνία προγραμματίζεται το 2020 να έχουν ε, και να λαμβάνουν 42% των συνολικών πληρωμών. Δεν είναι ικανοποιημένοι με το ποσοστό αυτό. Εσείς τι πιστεύετε ως ελεκτικό συνέδριο, οι άμεσες πληρωμές είναι δικές, ανταποκρίνονται στο πνεύμα της συνθήκης Λισαβόνας. Και μία δεύτερη ερώτηση. Ίσως να μην έχω ε, σαφή εντύπωση για την ε, έκταση, το εύρος των εργασιών σας, αλλά θα ήθελα να μάθω το εξής. Το Ελεκτικό συνέδριο λαμβάνει επιστολές, ε, αιτήματα από γεωργούς, από γεωργικές ενώσεις και αν λαμβάνει τέτοιες επιστολές, τι ζητούν να μάθουν το ελεκτικό συνέδριο οι και οι σχετικές ενώσεις. Ευχαριστούμε κύριε Ρούμπιξ. Η κυρία Μαγκίνη και μετά η κυρία Λούλινγκ. Μάρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ το ελεγκτικό συνέδριο για τη συνεισφορά τους εδώ σήμερα και για την έκθεση. Πάντα με απασχολεί κάτι από την προηγούμενη έκθεσή σας και θα ήθελα να αναφερθείτε σε αυτό το σημείο. Είναι στην παράγραφο 19 και αναφερθήκατε στην ε, πρώτη σας έκθεση για το σύστημα SPS. Ε, λέτε ότι η ενίσχυση προ γεωργού, οι οποίοι δεν είναι ενεργοί γεωργοί είναι διαδεδομένοι, αλλά δεν έχετε στοιχεία για να υποστηρίξετε αυτόν τον ισχυρισμό. Από πλευρά ελεγκτικού συνεδρίου ε, είναι περίεργη αυτή η δήλωση κατά την άποψή μου. Ε, κάνω παράφραση, αλλά αυτή είναι η ουσία αυτών που λέτε στην παράγραφο 19. Αν δεν το απαντήσετε τώρα, ίσω θα μπορέσετε να μου απαντήσετε στο μέλλον. Επίση, σε μια άλλη παράγραφο, την παράγραφο 12, που νομίζω ότι αναφέρει κάτι σημαντικό για το έργο μα εδώ, θα ήθελα να διευκρινίστε την ερμηνεία που δίνω στην παράγραφο 12. Λέτε ότι οι μεταρρυθμίσει, ακόμα και αν όλα πάνε καλά με τη δική μα τη δουλειά εδώ στο Κοινοβούλιο και με τα όσα θα κάνει το Συμβούλιο, θα ε, οδηγήσουν στο να χρειαστούν τα κράτη-μέλη 12 με 24 μήνες μετά από την έναρξη ισχύω ε, των κανονισμών για να δημιουργηθεί το σύστημα. Και αν όντω ισχύει αυτή η ερμηνεία που δίνω, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τις μεταρρυθμίσεις μέχρι την ημερημηνία που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνώ απολύτω ε, με τι ανησυχίε σα ε, για την απλούστευση και συμφωνεί και η Επιτροπή μας αυτό. Ίσως όμως ήρθε η ώρα να ρωτήσουμε το εξή μπορούμε να απλουστεύσουμε μια πολιτική που έχει μεταρρυθμιστεί τόσες πολλές φορές και σε αυτή τη σειρά των μεταρρυθμίσεων έχουμε και την πιο περίπλοκη ε, που είχαμε ποτέ διότι έχουμε αποσύνδεση από την παραγωγή. Ε, μπορούμε λοιπόν να το απλουστεύσουμε. Ίσως θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να δούμε τα πράγματα από άλλο πρίσμα. Διότι πολιτικός, αν ξανακούσω ακόμα μια φορά τον όρο απλούστευση, ακόμα και αν τον πω εγώ, μάλλον λάθος θα κάνω. Ε, κάνουμε κατάχρηση, ε, το υποσχόμαστε συνεχώς και δεν έχουμε ποτέ το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όσον αφορά τώρα το έτος αναφοράς, ε, το 2011-2014, νομίζω ότι κάνετε πολύ σημαντικές παρατηρήσεις που καλό θα ήταν να τις εξεργαστούμε και εμείς λίγο περαιτέρω. Για το κόστος, νομίζω ο παράγραφος 89, δεν κάνω λάθος, το κόστος για τους γεωργούς ε, προκειμένου να εφαρμόσουν τα μέτρα του greening. Εάν ακολουθήσουμε αυτή την άγουσα, θα πρέπει να υπάρχει ένα υπάλληλο τη Κομισιόν σε κάθε εκμετάλλευση για να δει ποιο κόστο δικαιολογείται και να αποφασίσει τι θα δίνεται και αυτό φυσικά θα περιπλέξει περισσότερο τα πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε άλλα μέσα προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο θα μας επιτρέψει να εργαστούμε. Ε, μπορείτε να δεχτείτε ότι όντως αυτό ισχύει και ποτέ δεν θα καταλήξουμε σε αυτή την ουτοπία που επιθυμούμε κι εσείς κι εγώ για τα σχόλιά σας για τον ενεργό ε, γεωργό νομίζω ότι είναι πολύ σωστή η οπτική σας και ίσως καλό θα ήταν να την ακολουθήσουμε και εμείς. Δεν ξέρω αν θα το δεχτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά υπάρχει ήδη ορισμό σε κάποιο κανονισμό και νομίζω ότι αν αλλάξουμε το ΜΕΙ με το ΣΑΛ θα διευκρινιστούν ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Για τον αρνητικό κατάλογο επίσης ε, μου κάνει νεύμα πρόεδρος να σταματήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκθεσή σας και θα ήθελα να μου απαντήσετε σε αυτά που σας ρωτώ. Ναι, έχουμε χρόνο, Μάριαν, μην ανησυχείτε. Έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Η κυρία Λούλινγκ και μετά ο Μάρτιν Χάουσλινγκ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω στον κύριο Κρέτα, το μέλος του ελεκτικού συνεδρίου, ότι έχω μείνει άναυδη. Είμαι χρόνια ολόκληρο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά δεν θυμάμαι ουδέποτε τέτοια συμπεριφορά του ελεγκτικού συνεδρίου. Φαίνεται να συμπεριφέρεται ο συνομοθέτης στο ελεγκτικό συνέδριο. Αυτό είναι άνω ποταμών και άνω προηγουμένου. Γιατί οι συνομοθέτες είναι μόνο το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποφασίσουν ε, πώ θα μεταρρυθμιστεί η κοινή γεωρική πολιτική, αν είναι χρήσιμη, ποιος είναι ο στόχος της κοινή γεωρικής πολιτικής. Από ό,τι ξέρω, δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ελεκτικού συνεδρίου ε, το θέμα των στόχων της ΚΑΠ, των σκοπών και των αποτελεσμάτων της και όλα αυτά που μας αναφέρετε. Μπορεί ρόλος του ελεκτικού συνεδρίου ε, να είναι οι οργανισμοί πληρωμών, οι οργανισμοί πιστοποίησης, αλλά δεν έχετε δικαίωμα όχι μόνο να μην να αποφασίσετε, αλλά ούτε να σχολιάζετε τους σκοπούς της κοινή γεωρικής πολιτικής και τους στόχους της. Αυτό είναι θέμα αρμοδιότητα των συνομοθετών. Μπορεί να, να ασκείτε κάποιο έλεγχο και να μας πείτε διάφορα θέματα ελεγκτικά, αλλά πού στηρίζεστε όταν λέτε ότι θέλετε να καθορίσετε τους στόχους της ΚΑΠ δεν είναι ρόλο αυτό και αρμοδιότητα του ελεκτικού συνεδρίου. Το ελεκτικό συνέδριο έχει ελεκτικό ρόλο. Δεν μπορεί να ανακατεύεται στη διαμόρφωση και το σχεδιασμό των πολιτικών. Αυτό δεν είναι δική σας δουλειά. Μπορείτε να συνεννοηθείτε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ελέξετε καλύτερα τους οργανισμούς πληρωμών και πιστοποίησης, πολύ ωραία, αλλά η διαμόρφωση και ο σχεδιασμός της πολιτικής αποτελεί αρμοδιότητα των συνομοθετών και όχι του ελεκτικού συνεδρίου. Ο κύριος Χόισλεν και μετά ο κύριος Δες. Yeah, Frage an den Μία ερώτηση προς το ελεκτικό συνέδριο συγκεκριμένη. Είπατε, χωρίς ε, ιδιαίτερα σχόλια, ότι η σημερινή μεταρρύθμιση θα σημαίνει 15% παραπάνω γραφειοκρατία. Αυτό το ελέγξατε εσείς ο ίδιος. Τι ελέγξατε ακριβώς και πώς ακριβώς προέκυψε αυτό το 15% γιατί εμένα μου φαίνεται κάπως σκοτεινό πώς είναι δυνατόν μια τόσο μικρή μεταρρύθμιση να έχει τόσο τεράστιο γραφειοκρατικό αντίκτυπο. Ίσως θα μπορούσατε να μου το εξηγήσετε. Εγώ δεν το κατάλαβα ούτε από αυτά που μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λίγο τώρα σε σχέση με αυτά που είπε και η κυρία Λούλινγκ. Αξιολογείτε και εκτιμάτε κάτι πολύ πολιτικό. Λέτε ότι η στοχοθέτηση δεν είναι δικαιολογημένη, δεν βλέπετε κάποιον συγκεκριμένη στοχοθέτηση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την οικολογική συνιστόσα. Μήπως κάπως υπερβαίνετε τις ερμοδιότητές σας έχετε στη διοίκησή σας ε, ανθρώπους που έχουν αργώνει, ασχοληθεί με θέματα, για παράδειγμα, βιοπικιλότητα στη γεωργία, θέματα προστασίας των υδάτων, του κλίματος. Είσαστε αρκετά απόλυτος, δεν νομίζω όμως ότι έχετε την αρμοδιότητα και την ικανότητα να κάνετε μια τεχνική πραγματικά αξιολόγηση του τι θέλει να πετύχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τη μείωση τη γραφειοκρατίας εν γέννη τώρα. Πάντα ε, το επικρίνετε κι εσείς, το επικρίνει κι άλλος κόσμος, ε, το σύστημα ελέγχου. Νομίζω ότι σε σχέση με τα 27 συστήματα των κρατών μελών μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν πολλά και διαφορετικά συστήματα ελέγχου. Και αν χρησιμοποιούσαμε εδώ το σύστημα των βέλτιστων πρακτικών, νομίζω ότι σε πολλές περιπτώσεις θα αποφεύγαμε πολλά στοιχεία της γραφειοκρατίας. γιατί θα βρίσκαμε τελικά ποιο σύστημα ελέγχου είναι το πιο αποδοτικό, το πιο αποτελεσματικό και το λιγότερο γραφειοκρατικό. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει πολλή γραφειοκρατία για την οποία δεν ευθυνόμαστε εμείς από τις Βρυξέλλες, αλλά τα κράτη-μέλη, τα κράτη αλλά πάντα κατηγορούνται οι Βρυξέλλες. Επειδή το είπε και η Μπρίτα Ράιμερς, ότι οι φτωχοί γεωργοί που τους υπερφορτώνουν διαρκώς με ελέγχους και τίποτα άλλο δεν έχουν να κάνουν παρά να ασχολούνται με τους ελέγχους. Θεωρείται ότι είναι υπερβολική η έλεγχη. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε αυτό και αν μιλάμε για τόσο μεγάλο ποσοστό χρηματοδότησης από τα δημόσια ταμεία, νομίζω ότι έχει δικαίωμα η δημόσια γνώμη να διεξάγει ελέγχους για να δικαιολογούνται αυτά τα ποσά. Ευχαριστώ ο κύριος Ντες και μετά Γιάρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Κροτάνα από το ε, ελεγκτικό συνέδριο για την παρουσίασή του. Μας ε, εξέπληξε κάπως ε, όπως τόνισαν και οι προλαλήσαντες. Αναρωτιέμαι κατά πόσον είναι έργο και καθήκον οποιοδήποτε ελεκτικού συνεδρίου της Βαυαρίας, της Γερμανίας, της Ευρώπης να αξιολογεί τέτοιους ε, γεωργικούς στόχους. Αυτό θεωρώ ότι αποτελεί ε, προνόμιο, δικαίωμα της πολιτικής. Γι' αυτό έχουμε εκλεχθεί εδώ από τους πολίτες. Δική σας, ε, δικό σας καθήκον είναι να διασφαλίζετε ότι η πρακτική αυτή και οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται λειτουργούν. Εκεί είμαι μαζί σας. Ο Ντόχρο Χέριν Κάιμερ θα ήταν σίγουρα ε, έκπληκτος ε, από το ελληνικό συνέδριο αν άκουγε αυτά που είπατε, γιατί δεν φαντάζομαι ότι σκόπευε να, ασχολη... να αναμειχθεί τόσο πολύ το ελεγκτικό συνέδριο στα της γεωργικής πολιτικής και σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις και τον έλεγχο της ορθότητας αυτών. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει ανάγκη να δράσουμε. Πολλές φορές το ακούσαμε και σήμερα ότι δεν γίνεται διάκριση στους ελέγχους κατά πόσον έγινε ένα λάθος, ένα σφάλμα ή κατά πόσον υπήρχε πρόθεση απάτης, εξαπάτησης. Γιατί κάπου μπορεί να γίνει ένα λάθος, το λάθος θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης, η απάτη μάλιστα να ε, συνεπάγεται κυρώσεις. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η διάκριση, γιατί πολλοί από το διοικητικό κλάδο μου λένε ότι ξέρουμε ότι ήταν λάθος και όχι πρόθεση, δεν υπήρξε πρόθεση εξαπάτησης, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να προβούμε σε κυρώσει, γιατί δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Κοινή αγροτική πολιτική, μήπως θα έπρεπε και αυτή η λέξη να ελεγχθεί, γιατί διαπιστώνω ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές στην Ευρώπη και ότι απέχουμε παρασάγκα από μια πραγματικά κοινή γεωργική πολιτική. Να δούμε, λοιπόν, τι γίνεται σε θέματα εφαρμογή και κατά πόσο τα κράτη-μέλη ανταποκρίνονται σε αυτήν την κοινή στοχοθέτηση για αυτό που είπατε για την πολλαπλή συμμόρφωση τώρα. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι σε θέματα πολλαπλή συμμόρφωσης διαπράξαμε ένα νομικό σφάλμα, θανάσιμο σφάλμα. Εγώ είμαι γεωργός, δεν είμαι νομικός. Δεν ξέρω γιατί λοιπόν ε, πουθενά αλλού στην Ευρώπη δεν υπάρχει διπλή ε, τιμωρία αν θέλετε παρά μόνο στην Γεωργία. Πουθενά αλλού δεν υπάρχει αυτό το σύστημα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει φυσικά επιβολή κυρώσεων, αλλά όχι διπλή. Και αυστηρές κυρώσεις, μάλιστα, αλλά όχι διπλές. Μια τελευταία ερώτηση. Θα μπορούσατε να μου πείτε ποιος ελέγχει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Onorevole ε, και μετά Λαβία. Να συμπληρώσω αυτό που είπε ο συνάδελφος. Είναι νομίζω αναμφίβολο ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ασχολείται με θέματα αποτελεσματικότητας των ε, κονδυλίων, των μέσων. Θα πρέπει να προσέξουμε γιατί η γραφειοκρατία δεν είναι, δεν και προκύπτει μόνο από την ε, διοικητική, το διοικητικό κλάδο, αλλά έχει και επιδράσεις και στη γεωργία. Και νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι υπηρεσίες ε, και παροχής πληρωμών δηλώνουν ότι δεν μπορούμε πλέον να τα βάλουμε πέρα. Και αυτό σχετίζεται με το πώς διασφαλίζουμε την αποτελεσματικότητα των κονδυλίων και πώς μπορούμε να τα διοχετεύσουμε τα κονδύλια αυτά στους γεωργούς. Νομίζω ότι στην σωστή κατεύθυνση κινούμαστε. Πώς μπορούμε λοιπόν να τα διαμορφώσουμε αυτά με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Είπατε ότι θα πρέπει να υπάρχει μία ε, γενική ευρωπαϊκή αρχή για την παροχή των κονδυλίων αυτών. Ναι, με, ναι, με αυτό θα έχει κάποια πλέον εκτήματα, αλλά πολύ φοβάμαι ότι αν υπήρχε μια τέτοια κεντρική αρχή θα ήταν ακόμα πιο μεγαλύτερη η γραφειοκρατία. Σε ό,τι αφορά τα διοικητικά αυτά έξοδα στα κράτη-μέλη, τα κράτη-μέλη πρέπει να προσέχουν ε, διπλά και τριπλά, γιατί σε περίπτωση οποιοδήποτε σφάλματος, είτε ήταν αυτό περιστασιακό, είτε ήταν ε, λόγω πρόθεσης, τελικά ε, επιβαρύνεται και είναι επιζήμιο το σφάλμα αυτό και για το γεωργό αλλά και για το κράτος μέλος. Πώς μπορούμε να μειώσουμε λοιπόν αυτό το άχθος και να ξέρουμε ότι υπάρχει και η πολιτική διάσταση. Λένε ότι οι συνάδελφοι, κάποιοι συνάδελφοι ότι είναι πολιτικά τα ζητήματα αυτά. Σας ρωτώ όμως και πάλι πώς μπορούμε να γίνει μια τέτοια μεταρρύθμιση με μικρό γραφειοκρατικό άχθος. Και μια άλλη ερώτηση που δεν έχει να κάνει μόνο με τη δική μου περιοχή σε ό,τι αφορά το κάπινγκ. Ανησυχώ ιδιαίτερα όταν οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τέτοια όρια. Με ανησυχεί το γεγονός ε, ότι στη Γερμανία διασπιστώνουμε ότι αυτό αφορά 30 επιχειρήσεις μόνο. Και τελικά η όλη αυτή ε, περίπλοκη γραφειοκρατική διαδικασία γίνεται για 30 επιχειρήσεις. Να μην χάνουμε δηλαδή από, το, από, από την ε, ε, τοπικό μας πεδίο και το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των μέτρων που λαμβάνουμε και να πάτε να το συνυπολογίζουμε το γραφειοκρατικό άχθος. Ευχαριστώ, Τζοβάνι Λαβία και μετά ο Τζιμ Νίκολς. E Νομίζω ότι από κάθε ανάγκη μπορούμε να βγάλουμε χρήσιμα στοιχεία για ε, τις δουλειές μας και νομίζω ότι η παρουσία του ελεγκτικού συνεδρίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επαληθεύσουμε και κάποια στοιχεία και της νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από την οπτική γωνία του ελεκτικού συνεδρίου και επομένω αυτού που κάνει το λογαριασμό. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τον εκπρόσωπο του ελεγκτικού συνεδρίου με στόχο να μειώσουμε αυτή τη μικρή διαφορά που, που υπάρχει μεταξύ του ηθελημένου σφάλματος, του ε, αθέλητου σφάλματος και της απάτης. Εάν το σύστημα το οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το greening και κυρίως στην περιτροπή καλλιέργεια και την ε, αγρανάπαυση ενός τμήματος ε, της έκτασης, αυτό το περιβόητο 7%. Επειδή σε αρκετές περιπτώσεις πρόκειται για πολύ μικρές ε, επιφάνειες, διότι μπορεί να είναι διαφορετική καλλιέργεια και στο εσωτερικό μιας εκμετάλλευσης πόσο περιθώριο αθέλου του σφάλματος μπορούμε να έχουμε, διότι σε μια μικρή επιφάνεια, ακόμα και 100 τετραγωνικών η διαφορά σε απόλυτες τιμές είναι το ίδιο, αλλά σε σχετικές τιμές για μια πολύ μικρή επιφάνεια μπορεί να είναι πολύ σημαντικό και επομένως ε, μπορεί να οδηγεί σε μια πολύ ε, στεναρή μετατόπιση που ε, είναι και αυτό το οποίο καθορίζει την κύρωση. Μήπως αυτό το στοιχείο λοιπόν ε, επηρεάζει αρνητικά τη δυνατότητα να κάνουμε σαφή διαχωρισμό μεταξύ του, ε, ενός ε, εκούσιου σφάλματος από την απάτη. Και θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Επειδή αναφερόμαστε συνεχώ στην απλούστευση και προσπαθούμε να προτείνουμε συνέχεια μέσα για την απλούστευση, θεωρείτε ότι κυρίω για τι ε, ε, μικρές επιχειρήσεις υπάρχει δυνατότητα να αξιολογήσουμε το ενδεχόμενο να κάνουμε κάποιες προτάσεις ε, πολιετής ε, κυρίως για τις ενισχύσεις ανεπιφάνεια ε, ιδίως όταν δεν υπάρχουν αλλαγές στην εκμετάλλευση και δεν υπάρχουν αλλαγές και στην υποδομή της εκμετάλλευσης να μπορούμε να τις έχουμε συνεχώς σταθερές χωρίς να υπάρχουν μεταβολές και να αποφύγουμε οι μικρές επιχειρήσεις να πρέπει κάθε χρόνο να κάνουν τις ίδιες αιτήσει, να αναπαράγουν την ίδια χαρτούρα και το ίδιο γραφειοκρατικό άκθος, το οποίο θα μπορούσε πολύ πιο εύκολα να ε, χρησιμοποιηθεί ε, στην ίδια την εκμετάλλευση, να μπορεί ο Γεωργός να διασπαταλήσει το χρόνο του στην εκμετάλλευσή του. Πόσο σημαντικό θεωρείται από πλευράς ελέγχου ότι θα πρέπει να παρουσιάζεται ε, κάθε φορά κάτι το οποίο να έχει συνέπειες, το οποίο να μην γίνεται μόνο για ένα χρόνο, αλλά να γίνεται για πολλά χρόνια. Δηλαδή, εάν δεν υπάρχει αλλαγή στην ακμετάλλευση, αν δεν αλλάγει ο παραγωγός φυσικά, αν δεν αλλάγει η μορφή της εκμετάλλευσης και να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο ε, μοντέλο για πολλά χρόνια. Ευχαριστώ, Τζοβάνι. Ο κατάλογος των ε, αγορητών κλείνει με τον Τζιμ Νίκολσον. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίσατε, ορίσατε, κύριε Κρετά. Νομίζω ότι συμφωνώ με τις ανησυχίες ε, ε κάποιον από την περιφέρεια μου. Είμαι δυόμιση χρόνια εδώ, δεν έχω ξαναδεί κάποιον από το ελεκτικό συνέδριο. Μπορεί να κάνω λάθος τουλάχιστον δεν μας είπε κανείς αυτά που μας είπατε εσείς σήμερα. Ίσως να αλλάζουν λοιπόν τα πράγματα και να ζούμε σε νέες εποχές. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τις απόψεις σας για το 15% ε, επιπλέον ε, του διοικητικού κόστους που θα έχουμε στον προϋπολογισμό, τι αίσθηση έχετε εσείς γι' αυτό. Και αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι ότι η Ευρώπη είναι μια πολυπίκυλη μεγάλη περιοχή από βορρά προς νότο, από ανατολάς προς τη μας. Ε, πολλές φορές πηγαίνω από τις Βρυξέλλες στο Στρασβούργο και κοιτάζω τους αγρούς όπως ε, οδηγώ και βλέπω ότι διαφέρουν πάρα πολύ από την ε, περιοχή μου στη Βόρεια Ιρλανδία όπου το ελεκτικό συνέδριο μας έδωσε πάμπολα εκατομμύρια πρόστιμο. Οι αγροί έγινε πολύ καιρό. Μπορεί να μην είστε εσείς ε, αυτοί οι οποίοι ήταν αρμόδιοι, αλλά κάποτε στο 16ο-17ο αιώνα υπήρχε χαρτογράφηση των αγρών και δεν καταλαβαίνω πώς ε, γίνεται να έχουμε τιμωρία για κάποιους και να μην έχουμε τιμωρία και για όσους ε, αλλάζουν τα πράγματα. Για να περάσω λοιπόν στην παρούσα κατάσταση και να σας πω πώς έχει η Ευρώπη σήμερα. Μπορούμε να συνεχίσουμε να υποχρεώνουμε συνεχώς ανθρώπους να εφαρμόζουν για όλα την ίδια λύση. Δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο απλούστευση γιατί δεν θέλω η Μάρια ε, να, ε, χάσει τη ψυχραιμία της, αλλά ε, κάπου πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση και θα πρέπει σε κάθε χώρα να υπάρχει ένας βαθμός ευελιξίας και να επιτρέπεται να υπάρχουν οι διαφορές ε, που υπάρχουν εντός της Ευρώπης και να έχουμε την καλύτερη χρήση ε, της κάθε εκμετάλλευσης όποτε μπορούμε να έχουμε τέτοιο. Ε, Κανένας δεν θέλει να έχει κατάχρηση κονδυλίων, κανένας δεν θέλει να το διαπιστώσει αυτό, αλλά φυσικά θα πρέπει να επιτρέψουμε και ένα βαθμό ευελιξίας. Και επιτρέψτε μου να πω, μην το πάρετε στραβά αυτό που θα σας πω, γιατί δεν ε, έχω κακή πρόθεση. Ίσως το γεγονός ότι είστε στο ελεκτικό συνέδριο δεν σας δίνει μια πλήρη εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει από αυτούς που προσπαθούν αφενός να εφαρμόσουν και ε, αφετέρου να διασφαλίσουν ότι εφαρμόζονται ορθώς οι κανόνες. Ελπίζω τις απόψεις μου να τις πάρετε ειλικρινά, διότι τα λέω με πάσα ειλικρίνεια και να τα λάβετε υπόψη, διότι είναι η πρώτη φορά που μου δόθηκε ευκαιρία να μιλήσω με μέλος του ελεκτικού συνεδρίου και πάντα είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι θα μιλήσω ευθέω και αυτό έκανα με σας και ελπίζω να τα κλάβετε έτσι και να μην θεωρήσετε ότι είχα κακή πρόθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο και τώρα πριν δώσω και πάλι το λόγο στο Μισελ Κρετάν να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπω το Διευθυντή τον κύριο Πατσέκο, παρακαλώ. Η Κομισιόν και μετά θα λάβετε εσείς το λόγο κύριε Κρετάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ε, Euh, Ευχαριστώ και τον κύριο Κρετά, το μέλο του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, για την παρουσίασή του. Φυσικά λαμβάνουμε πάντα σοβαρά υπόψη τι γνωμοδοτήσει του Ελεκτικού Συνεδρίου σε ό,τι αφορά τις πτυχέ τη χρηστή δημοσιονομική διαχείρισης και χαίρομαι που ε, το Ελεκτικό Συνέδριο αναγνώρισε τις προσπάθειες Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πολλού τομεί, γιατί δεν έχουμε μόνο κριτικέ και συστάσει. Σε πολλά σημεία το Ελεκτικό Συνέδριο αναγνωρίζει ε, την απλούστευση μέσα στις καλύτερες στόχευσης των ενισχύσεων, τη συγχώνευση ε, του μοντέλου με το καθεστώς ε, άμεσων πληρωμών και θεσπίσαμε ένα πλουστευμένο καθεστώς και για τους μικροκαλλιεργητές. Το ελεκτικό συνέδριο τάχθηκε υπέρ και των μέτρων που προτείνουμε για τους νέους γεωργούς, κάτι που δεν θα πρέπει επίσης να περάσει απαρατήρητο. Σε ό,τι αφορά τις παρατηρήσεις του του ελεκτικού συνεδρίου ε, για την περιπλοκότητα του καθεστώτος που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκαν τρία παραδείγματα. Το πρώτο, η ανάπτυξη της υπαίθρου. Θα έλεγα ότι έχουμε πια ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο που ισχύει για το σύνολο των διαρθρωτικών ταμείων, για όλα τα διαρθρωτικά ταμεία. Από εδώ και πέρα ε, η ανάπτυξη υπαίθρου θα γίνει σε ένα πιο συνεκτικό πλαίσιο και νομίζω ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό και αξιοσημείωτο. Σε ό,τι αφορά την οικοαιρεσιμότητα, έχει μειωθεί ο αριθμός των προϋποθέσεων και των απαιτήσεων, κάτι που αποτελεί απλούστευση. Αλλά έχουμε και πολλούς στόχους ε, που εξυπηρετεί η οικοαιρεσιμότητα. Δεν μπορούμε να τους υλοποιήσουμε χωρίς να προβλέψουμε αρκετά κριτήρια και κανόνες. Ό,τι αφορά τις κυρώσεις, συμφωνώ με τις απόψεις ε, των πολλών ευρωβουλευτών και του κυρίου Ντές. Το θέμα της οικοαιρεσιμότητας δεν είναι θέμα επιλεξιμότητας. Δεν πρόκειται δηλαδή να πλήξουμε το σύνολο της ενίσχυσης ε, που λαμβάνει ο Γιώργος. Μόνο σε περίπτωση που δεν τηρούνται κάποιοι κανόνες ε, θα υφίσταται κυρώσεις ο Γιώργος. Ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι αυτό των ενεργών γεωργών. Πιστεύω και δεν είμαστε αυτιστικοί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν αμφαλοσκοπούμε. Ακούσαμε με ιδιαίτερη προσοχή τις επικρίσεις ε, για τις προτάσεις μας. Εμείς προτείνουμε μόνο οι πραγματικοί γεωργοί, ενεργοί γεωργοί να δικαιούνται άμεσες πληρωμές. Νομίζω ότι δεν μπορεί να διαφωνήσει α, κανείς γι' αυτό, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε η Επιτροπή Γεωργίας, ούτε το Ελεκτικό Συνέδριο. Καταθέσαμε λοιπόν κάποιες προτάσεις που επικρίθηκαν ως υπερβολικά περίπλοκες, πολυσύνθετες και ε, γραφειοκρατικές. Μια και σαν το εθνικό γραφειοκρατικό άχθος. Προτείναμε λοιπόν να να έχουμε ένα θετικό ορισμό, να έχουμε έναν αρνητικό ορισμό, έναν αρνητικό κατάλογο. Και νομίζω ότι λάβαμε υπόψη και δικές σας προτάσεις με τον αρνητικό κατάλογο. Ε, όσοι περιλαμβάνονται σε αυτό το κατάλογο, σε περίπτωση που θεωρούν ότι είναι ε, γεωργικές επιχειρήσεις, εναπόκειται σε αυτούς να αποδείξουν ότι όντως είναι ένεργοι γεωργοί. Και έτσι μειώνεται σημαντικά το γραφειοκρατικό άκθος και των εθνικών διοικήσεων. Αντί να γίνεται προκαταρκτικός έλεγχος όλων των αιτήσεων, θα γίνεται μία επαλήθευση μόνο σε περίπτωση που κάποιος που περιλαμβάνονται στον αρνητικό κατάλογο ισχυρίζεται ότι είναι επιλέξιμος, ότι εμπίπτει στον ορισμό του ενεργού Γιώργου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο πλούστευσης. Άλλο θέμα το, της κατανομής των ενισχύσεων. Η κυρία Μαγκίνες απάντησε ξεκάθαρα στην ερώτηση αυτή. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Ασθενίζομαι πλήρω στην απάντηση της κυρίας Μαγκίνες. Σε ό,τι αφορά τους οργανισμούς πληρωμής, θεωρούμε ότι έχουμε εδώ μεικτή διαχείριση, κοινή διαχείριση, επιμερισμένη με τα κράτη-μέλη. Οπότε και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμβάλλουν σε αυτή τη διαχείριση. Εμείς κάνουμε ένα δειγματοληπτικό έλεγχο, ετήσιο, για να εξακριβώσουμε πώς ε, ε, εργάζονται οι οργανισμοί πληρωμής. Αν κατά τη γνώμη μας υπάρχουν αποκλήσεις ως προς τον ε, δημοσιονομικό κανονισμό, θα το λάβουμε υπόψη και θα ενεργήσουμε αντίστοιχα. Θεωρούμε ότι αυτό το σύστημα έχει αποδείξει τη λειτουργικότητά του και υπάρχουν και πολλές βελτιώσεις. Αυτά προς το παρόν κύριε Πρόεδρε για την έκθεση του Ενεκτικού Συνεδρίου την οποία θα εξετάσουμε με ιδιαίτερη προσοχή και είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις. Ευχαριστώ πολύ τον ε, κύριο Πατσέκο. Και τώρα δεν υπάρχουν άλλοι που ζητούν το λόγο, να δώσουμε το λόγο στο Μισελ Κρετά. Και πάλι σας ευχαριστώ για τη σημερινή σας παρουσία εδώ και γιατί μας παρουσιάσατε την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, θα το προσπαθήσω πάντως. Καταρχήν μια ερώτηση που ε, διατυπώθηκε επανειλημμένος. Να δώσω κάποιες γενικές εξηγήσεις ως προς τις πολιτικές επικρίσεις που έγιναν. Κατά πόσο το ελεκτικό συνέδριο χαράζει την κοινή γεωργική πολιτική. Η απάντηση είναι αρνητική φυσικά. Ουδέποτε δεν είχαμε την πρόθεση να αντικαταστήσουμε την Επιτροπή στο Δικαίωμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας της ή το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο στις νομοθετικές τους αρμοδιότητες και στην αρμοδιότητα καθορισμού και έγκρισης της κοινωτικής νομοθεσίας. Αλλά καλούμαστε να δώσουμε τη γνώμη μας για διάφορα θέματα. Μα προσάψετε ότι θέλουμε να προσδιορίσουμε του στόχου τη κοινή γεωργική πολιτική. Λάθο, καθόλου. Μπορεί εγώ να μην ε, εκφράστηκα σωστά, αλλά ουδέποτε δεν έδωσα κάποιους προσιορατολισμούς του ελεκτικού συνεδρίου για την ακολουθητέα κατεύθυνση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Είπα όμως ότι χωρίς στόχους είναι δύσκολο να αποτιμήσουμε τα αποτελέσματα. Δεν είπα ποιοι θα πρέπει να είναι οι στόχοι της κοινή γεωργικής πολιτικής. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα προηγουμένως. Κοιτάξτε τον κανονισμό για τις άμεσες πληρωμές. Και πείτε μου, βλέπετε πουθενά στον κανονισμό αυτό να προσδιορίζονται στόχοι πουθενά στον κανονισμό δεν αναφέρονται στόχοι. Δεν είπα εγώ ποιοι θα πρέπει να είναι οι στόχοι. Είπα απλώ ότι λείπουν οι στόχοι από τον κανονισμό. Το ίδιο και για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Εκεί είχαμε αντίστροφη κατάσταση. Εκεί έχουμε χίλιους στόχους, ένα σωρό στόχους έχουμε μια μισή σελίδα, ένα μακροσκελέστατο κατάλογο με απαρίθμιση των στόχων. Μερικοί μάλιστα είναι και αντιφατικοί μεταξύ τους, άλλοι είναι συγκεχημένοι, άλλοι είναι αόριστοι. Είπα ότι για την ανάπτυξη της υπαίθρου θα πρέπει να απλοποιηθούν, να απλουστευθούν οι στόχοι, να γίνει καλύτερη στόχευσή τους, καλύτερη εστίασή τους τη διευκρίνηση. Δεν είπα όμως ποιοι θα πρέπει να είναι αυτοί οι στόχοι αρνούμε κατηγορηματικά τις κατηγορίες εντός εισαγωγικών, τις μορφές που ασκήθηκαν κατά του ελεκτικού συνεδρίου, ότι θέλουμε να παρεύουμε σε τομέα που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα μας, επουδενή. Απλώς, επειδή το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο έχει δικαίωμα να γνωμοδοτήσει ως του προ τι ε, βασικέ προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεμελιώδει προτάσει που έχουν δημοσιονομικέ επιπτώσει και να παρουσιάσει αυτή τη γνώμη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό κάνουμε. Υποβάλλουμε αυτή την έκθεση που είναι η γνωμοδότηση του Ελεκτικού Συνεδρίου που υποβάλλουμε στην Επιτροπή Γεωργία και στην Επιτροπή Προπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ω προ τι δημοσιονομικέ επιπτώσει κάποιων νομοθετικών προτάσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για παράδειγμα, δεν έχω καμία απάντηση προς τον κύριο Ρούμπιξ που με ρώτησε αν κρίνω ότι οι χαμηλότερες πληρωμές που έγιναν στους Λετωνούς ε, γεωργούς ήταν δικαιολογημένες ή όχι. Εγώ δικαιούμαι να εξακριβώσω κατά πόσο ο υπολογισμός των πληρωμών συνάδει με τις κοινοτικές διατάξεις και αν είναι νομότυπος. Δεν πρόκειται να κρίνω τη σκοπιμότητα ή το ύψος αυτών των πληρωμών σε καμία περίπτωση δεν εξέφερα πολιτική γνώμη για το τι χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει η κοινή γεωρική πολιτική. Απλώ είπα ότι για να μπορέσουμε να αποτιμήσουμε και να καταμετρήσουμε τα αποτελέσματα τη κοινή γεωρική πολιτική, χρειαζόμαστε στόχου και δείκτε για να κάνουμε έναν απολογισμό των αποτελεσμάτων. Και είπα ότι ούτε δείκτε αποτελεσμάτων υπάρχουν στου κανονισμού, ούτε στόχοι. Ένα δεύτερο λάθος που θα ήθελα να διορθώσω και μια ανησυχία να διασκεδάσω. Διαφορά μεταξύ ε, εκούσιου ή ακούσιου σφάλματος και απάτης. Μπορεί να σας απογοητεύσω, αλλά για το ελεκτικό συνέδριο δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ εκούσιου σφάλματος και απάτης. Το ελεκτικό συνέδριο ούτε δικαίωμα έχει, αλλά ούτε και στόχο έχει να διώξει τους απαταιώνες. Δεν είναι το ελεκτικό συνέδριο αυτό που διώκει τους διαπράδοντες ατασταλίες. Αν απλώς στη διάρκεια των ελέγχων διαπιστώνουμε κάποιες απάτες, φέρουμε την ευθύνη να κοινοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία που στοιχειοθετούν απάτη ή υποτιθέμενη απάτη, υποχρεούμαστε να διαβιβάσουμε αυτά τα στοιχεία στα εθνικά δικαστήρια. Το ελεγκτικό συνέδριο δεν είναι δικαστήριο, δεν ελέγχει, ούτε ασκεί διώξει για απάτες, ούτε κάνει διάκριση μεταξύ των εκούσεων ή ακούσεων σφαλμάτων. Το ελεγκτικό συνέδριο υποβάλλει μια αντικειμενική κρίση για το γεγονός ότι κάποιο ποσό, κάποια δαπάνη επιρρήθηκε στον κοινοτικό προϋπολογισμό αδικαιολόγητα. Δεν ενδιαφέρεται το ελεκτικό δικαστήριο για ποιο λόγο έγινε αυτή η ατασταλία και για αυτό λόγο παράτυπα μια συγκεκριμένη δαπάνη ε, περιλήφθηκε στον κοινοτικό προπολογισμό. Μα ενδιαφέρει το γεγονό απλώ ότι αχρεώσετα καταβλήθηκε μια δαπάνη. Δεν, γίνεται για μας, δεν υπάρχει διάκριση για μα μεταξύ σφάλματο και απάτη. Από τη στιγμή που εντοπίζουμε κάποια απάτη, διόλια συμπεριφορά, κοινοποιούμε τα στοιχεία, διαβιβάζουμε τα στοιχεία στην ε, στα εθνικά δικαστήρια. Δεν πρόκειται εμεί να απαγγείλουμε κατηγορίε ή να βρούμε ποιο είναι ο υπέτειο. Απλώ διαπιστώνουμε κατά πόσο ε, οι λογαριασμοί, το ύψος των δαπανών που υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο, αυτό το ύψος ε, των δαπανών είναι νομότυπο ή όχι, ή αν υπάρχουν ατασταλίε. Αυτό μόνο εξακριβώνει το ελεκτικό συνέδριο. Και να απαντήσω παρεπιπτόντως και στον κύριο Νίκολσον. Το ελεκτικό συνέδριο ουδέποτε δεν επέβαλε ε, στην Βόρεια Ιρλανδία πρόστιμο 120 εκατομμυρίων, εκατομμυρίων λιρών στερελίνων. Δεν έχει τέτοιο, τέτοια αρμοδιότητα το ελεκτικό συνέδριο, ούτε δικαίωμα ούτε εξουσία. Είναι αδύνατον το ελεκτικό συνέδριο να επέβαλε πρόστιμο 120 εκατομμυρίων λιρών στη Βόρεια Ιρλανδία. Μπορεί να αναφέρεστε σε μια διόρθωση αλλά σε καμία περίπτωση αυτό δεν είναι πρόστιμο που επευλήθη από το ελεκτικό συνέδριο στη Βόρεια Ιρλανδία, γιατί δεν δικαιούται να κάνει κάτι τέτοιο το ελεκτικό συνέδριο. Μετά τις διευκρινήσεις λοιπόν αυτές θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ορισμένες ερωτήσεις. Με τη σειρά που διατυπώθηκα στο μέτρο του δυνατού. Κυρία Κέστιγκερ, ρωτήσατε μήπως αν ε, αιτία της ε, πολυπλοκότητας ε, της γεωργικής ομοθεσίας πηγάζει και από τα κράτη-μέλη. Η απάντηση είναι θετική, καταφατική. Το κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο αφήνει ένα περιθώριο λιγμό στα κράτη-μέλη, αφήνει μια ευχέρεια εκτίμησης στα κράτη-μέλη για να προσαρμόσουν τη γενική νομοθεσία στις ιδιαίτερες συνθήκες τους. Και απαντώ έτσι και στον κύριο Νίκολσον που υπέβαλε παρόμοια ερώτηση. Αν μπορεί ένας, ο, ο ίδιος κανόνας να ισχύει για όλους. Όχι, ε, ένας κανόνας δεν ισχύει για όλους. Για παράδειγμα, στα, στην οικοαιρεσιμότητα έχουμε δύο κατηγορίες προϋποθέσεων. έχουμε τα statutory management requirements που λέμε στα αγγλικά και το από την άλλη πλευρά της good agricultural and environmental conditions. Η δεύτερη κατηγορία καθορίζεται σε επίπεδο κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη καθορίζουν τις σωστές περιβαλλοντικές και γεωργικές συνθήκες, όχι, τα, όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε και τα κράτη-μέλη μπορεί να συμβάλλουν σε αυτή την περιπλοκότητα. Για παράδειγμα, τα κράτη-μέλη δίνανται, ορίζοντα αυτές τις περιβαλλοντικές και, γεωργικέ συνθήκε να περιπλέξουν τις απαιτήσει ε, της οικοαιρεσιμότητα. Άρα και αυτά είναι συνυπεύθυνα για την πολυπλοκότητα που έχει δημιουργηθεί. Υπάρχει μία αυτονομία, ένα περιθώριο λιγμών των κρατών μελών στην προσπάθεια ε, Προσαρμογή τη γενική νομοθεσία στις ε, εθνικές ιδιαίτερότητε. Στην περίπτωση των ΚΑΕΓ, της οικοαιρεσιμότητας σε ό,τι αφορά τι περιβαλλοντικέ συνθήκε. Ε, αρμόδια για τον καθορισμό τους είναι τα κράτη-μέλη. Και η περιπλοκότητα της διαχείρισης ε, οφείλεται εν μέρη στο γεγονό ότι τα κράτη-μέλη προσθέτουν κάποιες εθνικές νομοθετικές διατάξεις στις κοινοτικέ νομοθετικές διατάξεις και έτσι επιτείνεται η πολυπλοκότητα. Αλλά όταν είπε το ελεγκτικό συνέδριο ότι η, η γεωργική νομοθεσία είναι πολύ σύνθετη. Δεν είχαμε αυτό στο μυαλό μας, δηλαδή την προσθήκη των, των νομοθετικών διατάξεων εκ μέρου των κρατών μελών. Ναι, μεν είναι ένα στοιχείο τη περιπλοκότητα αυτή η προσθήκη, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Για την ανάπτυξη τη υπαίθρου, όπω σα είπα, έχουμε έξι στρώματα νομοθεσία. Η εθνική νομοθεσία είναι το έκτο στρώμα. Προηγούνται άλλα πέντε στρώματα. που είναι κοινοτική προέλευση. Και εκεί θα μπορούσαν να γίνουν απλοποίησει λοιπόν. Το θέμα της απλούστευσης δεν είναι τόσο εύκολο στην ανάλυση, γιατί υπάρχουν και καλές απλουστεύσεις και χειρότερες. Στην περίπτωση της οικοαιρεσιμότητας, δεν μπορούμε να έχουμε διατάξεις για την οικοαιρεσιμότητα γενικές και όριζες. Πρέπει να είναι κάπως πιο λεπτομεριακές να είναι πιο ενδελεχείς, να μιλούν το καθεστώς χρήσης του ύδατος, διαφύλαξη του εδάφους, συντήρηση του εδάφους, το ποσοστό των ε, ε, αζωτούχων στα λοιπάσματα, ε, λύματα λίματα με υψηλή περιεκτικότητα σε αζωτούχες ενώσεις. Δεν μπορούν να είναι αυτά όλα γενικά ούτε απλά, γιατί όντω, η κατάσταση είναι περίπλοκη. Θα πρέπει να υπάρχει ένα βαθμό λεπτομέρειε. Για να απλουστευτούν όμω τα πράγματα θα πρέπει να εξηγήσουμε καλά την κατάσταση στου γεωργού. ώστε να γνωρίζουν οι γεωργοί όταν δεσμεύονται για την οικορεσιμότητα, τι προϋποθέτει αυτή. Βέβαια, ένα τμήμα της οικορεσιμότητας είναι υποχρεωτικό για όλους, αλλά υπάρχει και ένα τμήμα, όπως τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα που είναι προαιρετικά. Θα πρέπει λοιπόν να έχουν γνώση οι γεωργοί γιατί δεσμεύονται. Πάντως πρόκειται για ένα σύνθετο, πολυσύνθετο σύνολο που δεν πρόκειται να απλουστευτεί διαμαγίας. Γιατί είναι περίπλοκο το θέμα, λογικό είναι και οι διατάξεις σύνθετες. Σήμερα για παράδειγμα τα SMA απορρέουν από 18 διαφορετικά νομοθετικά κείμενα. Ίσως ένα μέτρο απλοποίησης θα ήταν μία αναδιατύπωση και μία οργάνωση με συγκροτημένο τρόπο ανά τομέα. Ένα τομέα στο είδωρο, άλλο τομέα στο έδαφο, τρίτο στα λοιπάσματα και ούτω καθεξής. Και αντί να έχουμε 18 διαφορετικά νομοθετικά κείμενα, στο οποίο πρέπει να ανατρέξει κανείς για να βρει τα SMA, μπορεί ε, όλα αυτά να συμπεριληφθούν σε ένα ενιαίο και συνεκτικό κανονιστικό πλαίσιο. Αυτό θα ήταν ένα μέτρο απλούστευσης. Συμβατό όμως με τον απαραίτητο βαθμό λεπτομέρειας που απαιτείται. το greening, το πρασίνισμα θα πρέπει να εμπίπτει στον πρώτο ή στο δεύτερο πυλώνα. Τι να σου πω, αυτά είναι πολιτικά ζητήματα. Δεν έχω αρμοδιότητα. Δεν δικαιούται το ελεκτικό συνέδριο να αποφασίσει αν το πρασίνισμα θα πρέπει να εμπίπτει στα μέτρα του πρώτου ή του δεύτερου πυλώνα. Σήμερα ένα τμήμα των μέτρων του πρασινίσματος περιλαμβάνονται στο πρώτο πυλώνα, ισχύουν για όλους και υπάρχουν και ειδικά μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο των σχεδίων ανάπτυξη πέθρου, στα πλαίσια των αγροπεριβαλλοντικών συμβάσεων και άρα εμπίπτουν στο δεύτερο πυλώνα. Υπάρχει ένας καταμερισμός των μέτρων πρασινίσματος μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα. Πάντως, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι και πολύ λογικό να έχουμε ένα κοινό βάθρο πρασινίσματος που θα ισχύει για όλους, άσχετα με την περιοχή και την δραστηριότητά τους. Και μετά να έχουμε ένα δεύτερο στοιχείο πρασινίσματος, πιο απαιτητικό και μάλιστα θα επιβραβεύεται με επιχορηγήσεις και αποτελεί κατά το αντικείμενο των συμβάσεων. Αυτό είναι στο δεύτερο πυλώνα. Υπάρχει ένας καταμερισμός η ισορροπία μεταξύ του υποχρεωτικού γενικής εφαρμογής μέτρου και του προαιρετικού μέτρου που επιβραβεύεται με επιχορηγήσεις ε, δεν είναι κατά κακή. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο για αυτό το θέμα. Υπάρχει και μια συσσόρευση των ελέγχων και μάλιστα σε ένα μόσποδο υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη επικάλυψη γιατί έχουμε και τους ε, ελέγχους των κρατηδίων που ε, προστίθενται στους ε, κεντρικούς ομοσπονδιακούς ελέγχους, έχουμε επιπλέον τους ελέγχους Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά και τους ελέγχους του Ελεκτικού Συνεδρίου. Οπότε μπορεί ο ίδιος Γεωργός να δει να περάνε τα μάτια του πέντε διαφορετικά ελεκτικά επιτελεία, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Θεωρητική είναι αυτή η πιθανότητα, αλλά είναι αλήθεια ότι υπάρχει ε, μεγάλη συσσόρευση ελέγχων. Αλλά δεν έχω μέτρα να προτείνω. Θα μπορούσαμε να μειώσουμε τους ελέγχους αν κάθε ε, επίπεδο ελέγχου μπορεί να στηριχθεί στους προηγούμενους ελέγχους που έγιναν σε χαμηλότερο επίπεδο. Αν ήμασταν σίγουροι για την ορθότητα των ελέγχων, αν πούμε το ελεκτικό συνέδριο ήταν βέβαιο ότι η έλεγχη των οργανισμών πιστοποίησης είναι σωστή και αξιόπιστη, θα μπορούσαμε να τους θεωρήσουμε ως δεδομένους, να στηριχθούμε σε αυτούς και απλώς να, να εξακριβώσουμε τη σωστή του λειτουργία και να αισθενιστούμε τα πορίσματα των ελέγχων τους, να μην χρειαστεί να τους επαναλάβουμε. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες προτάσεις, αλλά δεν έχει απλοποιηθεί πλήρως αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, Κυρία Μαγκίνης, πρέπει να σας πω ότι δεν κατάλαβα απόλυτα καλά την ερώτησή σας. Είπατε ε, Καταρχάς κάτι για την παράγραφο 12 της γνωμοδότησής μας, αν ε, κατάλαβα καλά. Α, το θέμα του χρόνου προσαρμογής ε, των ε, εκμεταλλεύσεων. Ναι, πράγματι θεωρούμε ότι οι οργανισμοί πληρωμών θα πρέπει Το πλήρες καθεστώς στο οποίο θα υπόκεινται θα είναι γνωστό. Αυτή τη στιγμή θα εφαρμόζεται ο κανονισμός. Και αυτή τη στιγμή οι εφαρμοστικές ε, πράξεις, οι εκτελεστικές πράξεις θα προχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην έχουν αρκετό χρόνο οι οργανισμοί πληρωμή για να ε, προσαρμοστούν και μπορεί να πρέπει να πάνε πέρα από το τέλος του 2013 για να μπορέσουν να εφαρμόσουν το νέο κανονισμό. Όντως υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Επειδή ε, ε, είμαι σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να φέρω κάτι για αυτό το 15%. Κάποιος με ρώτησε κατά πόσον γνωρίζω τι περιλαμβάνει, ε, αν επαληθεύθηκε αυτό το, από το ελεκτικό συνέδριο. Αυτό με ρωτήσατε, αν το 15% επαληθεύθηκε από το ελεκτικό συνέδριο. Όχι, δεν έχει επαληθευθεί από το ελεκτικό συνέδριο. Το 15% είναι το ποσοστό που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις επιπτώσεις της νομοθεσίας. Μεταξύ λοιπόν των εγγράφων που σας έχει υποβάλει, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει και μία εκτίμηση των ε, δημοσιονομικών επιπτώσεων αυτό που προτείνει και έχει ε, εκτιμήσει ότι περίπου 15% του παρόντος κόστους διαχείρισης θα είναι επιπλέον. Επειδή δεν υπάρχει κάποια απάντηση για αυτό το νέο καθιστώ, το ελεγκτικό συνέδριο δεν έχει κάνει επαλήθευση δαπανών. Θα το κάνουμε το 2014, το 2015 ή το 2016. Αλλά είναι σαφές του, του λεχθέντος ότι το νέο καθεστώς περιλαμβάνει και κάποιες επιπλέον δαπάνες. Ε, ένα παράδειγμα να σας δώσω μόνο. Εάν οι οργανισμοί πιστοποίησης πρέπει όχι μόνο να εκφράσουν την άποψή τους για τη βιωσιμότητα των λογαριασμών, αλλά και για την ομιμότητα και την ε, ε, ομαλότητα των συναλλαγών, τότε θα χρειάζεται πολύ περισσότερο προσωπικό, θα χρειάζεται πολύ περισσότερη εργασία και επομένως θα κοστίζει περισσότερο. Δεν μπορώ να δω πώς θα μπορέσουμε να έχουμε λιγότερες δαπάνες. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος, αλλά σίγουρα θα στοιχίζει ακριβότερα διότι θα έχουμε πιο σημαντικά καθήκοντα. Η παράγραφος 19 τώρα. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν είχα καταλάβει καλά. Είχα σημειώσει 9. Λοιπόν, τι λέει η παράγραφος αυτή. Η 19. Α, η 90, συγγνώμη, η 90. 9-0. Παρακαλώ. Η κυρία Μακίνες, Ίσως θα μπορούσατε να μου γράψετε την απάντηση. Μου φαίνεται πολύ περίεργο ότι ένας ελεγκτής, γιατί σχεδόν ήμουν κι εγώ ελεγκτής, να λέει ότι το πρόβλημα είναι πολύ διαδεδομένο, αλλά λέει ότι ούτε τα κράτη-μέλη που επισκεφθήκαμε, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ακριβεί πληροφορίε για αυτό το φαινόμενο που λέτε ότι είναι πολύ διαδεδομένο. Πώ μπορείτε να κάνετε τέτοια δήλωση νομίζω ότι την έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση. Μπορούμε να κάνουμε τη δήλωση, διότι κάθε χρόνο επισκεφτόμαστε ένα μεγάλο αριθμό κρατών μελών, πηγαίνουμε σε πολλές εκμεταλλεύσεις και δεν είναι κάτι το οποίο το διαπιστώνουμε από καιρού καιρών ουσιαστικά σε όλα τα κράτη-μέλη που επισκεφθήκαμε, σε κάθε, ίσως όχι σε κάθε εκμετάλλευση, αλλά σε πολλές από τις εκμεταλλεύσεις που πήγαμε, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν αρκετά παραδείγματα και υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία, δεν τα έχω εδώ, αλλά έχουμε δημοσιεύσει μια συγκεκριμένη έκθεση όπου υπάρχει ένας μακροσκελέστατος κατάλογος όλων αυτών των παραδειγμάτων δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω εδώ, αλλά σας είπα, αεροδρόμια, ε, σιδηροδρομικές εταιρείες, κλαμπ ε, γκολφ, ε, ε, φυσικοί βιότοποι, ε, χώροι ψυχαγωγίας και αθλητισμού και ούτω καθεξής. Και αυτά τα έχουμε διαπιστώσει ολούθε. Σας λέω λοιπόν ότι είναι διαδεδομένο. Τώρα, δεν μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε αυτή τη δήλωση. Δεν έχουμε τους πόρους για να το κάνουμε, αλλά ε, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε τη δήλωση. Να σταματήσω εδώ νομίζω, ε. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Μισελ Κρετάν. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Και σε αυτό το σημείο, δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, νομίζω ότι περατώθηκε αυτό το διήμερο συνεδρίασης. Ε, σας ξαναδίνουμε ραντεβού για τις 8 Μαΐου στις 3 η ώρα και θα ήθελα να ζητήσω από τους συντονιστές και τους εισηγητές να παραμείνουν, διότι αμέσως μετά θα κάνουμε μια συνεδρία συνεδρίαση συντονιστών. Ευχαριστώ όλους και θα τα ξαναπούμε στις 8 Μαΐου και ευχαριστούμε και το ελεκτικό συνέδριο. Merci beaucoup. Très, gentil et très